Dear colleagues, please, Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ. Ας προχωρήσουμε στην έγκριση της ημερησίας διάταξης. Εγκρίνεται. Και καλωσορίζω τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τον κύριο Μάριο Ντράγκη, για το πρώτο νομισματικό διάλογο του νέου έτους. Ο προηγούμενο θα θυμάστε είχε λάβει χώρα στις 28 Νοεμβρίου. Ο σημερινό λαμβάνει χώρα σε μια συγκυρία περίπλοκη, γεμάτη προκλήσεις. Βλέπουμε τα οικονομικά δεδομένα μένα, αλλά παραμένουν αρνητικές οι προβλέψεις για την Ευρωζώνη λόγω των γεωπολιτικών παραγόντων κυρίως και κυρίως ε, συγκεκριμένα επιβεβαίωσης μονομερών επιλογών της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών, κυρίως όσον αφορά ζητήματα ρύθμισης των χρηματοπιστωτικών αγορών. Όλα αυτά γεννούν ανησυχίες, απαιτούν διεξοδική μελέτη και δράση από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας εκ τούτου, η διαφοροποιημένη ολοκλήρωση μπορεί και οφείλει να καταστεί σημαντικό εργαλείο, αλλά μέσα στο πλαίσιο του νέου, ε, της νέας ένωμης τάξης και της διατήρησης ε, της συνοχής της Ευρωζώνης και της δυνατότητάς της για την επίτευξη ε, των φιλοδόξων στόχων, δηλαδή της ολοκλήρωσης της ΟΝΕ, ποτέ προς την αντίθετη κατεύθυνση. Η στάση της ΕΚΤ, όπως γνωρίζετε, πάντοτε ήταν ε, αμετακίνητη, συνεχίζει την αγορά το πρόγραμμα αγοράς τίτλων από το 2000, έως το 2017 με ρυθμούς ε, της τάξης των 60 δισεκατομμυρίων μέχρι το Δεκέμβριο του 2017 και ή ε, εάν καταστεί απαραίτητο μπορεί να συνεχίσει και περαιτέρω, εν πάση περιπτώσει όσο χρειαστεί για την επίτευξη ενός ε, στόχου πληθωρισμού. Το μήνυμα λοιπόν της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι ότι δεν θα επιτρέψει να ε, τεθεί ένα αμφιβόλο η μετριοπαθής αλλά σταθερή ανάπτυξη της Ευρωζώνης και ότι έχει επαρκή ε, όπλα στη διάθεσή της, επαρκή μέσα στη διάθεσή της για να εξασφαλίσει τους στόχους αυτούς. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική τράπεζα έχει με, τους, ε, με, τους, ε, με τις πολιτικές της, ε, τις μη συμβατικές πολιτικές θα δραματίσει κέριο ρόλο, έχει εξασφαλίσει σταθερότητα τιμών και αγορών. Υπάρχουν κάποιες ανησυχίες σε σχέση με ενδεχόμενες αντίξωες συνέπειες των νομισματικών πολιτικών, των πρόσθετο κίνδυνο, παραδείγματι, σε σχέση με την χρηματοοικονομική σταθερότητα από το πρόγραμμα της, ε, νομίζω, της προσωπικής χαλάρωσης, ζητήματα μεταξύ άλλων που έχουν απασχολήσει και τους συντονιστές της Επιτροπής των Οικονομικών μας εν ώψη της προετοιμασίας για τον νομισματικό διάλογο, που αναπτύχθηκε βεβαίως σε συνεργασία και με διακεκριμένους καθηγητές με μια πρώτη έκθεση η οποία δείχνει πως τα στοιχεία δεν δίνουν σαφή αντίληψη συνένεσης ως προς την δημιουργία πιθανών, ε, πιθανής φούσκας από το σύστημα προσωπικής χαλάρωσης. Όσον αφορά δε τα άλλα ζητήματα, η μελέτη αποδικ... Ε, σημειώνει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία πως η νομισματική πολιτική μπορεί να έχει επηρεάσει την παραγωγικότητα. Πολλά και ενδιαφέροντα τα θέματα που έχουμε να συζητήσουμε. Πολλές οι προσδοκίες από την δική σας ομιλία, Πρόεδρε Τράγκη, και σας δίνω το λόγο. Thank Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμοι ε, Ευρωβουλευτέ, μέλη της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων. Κυρίες και κύριοι, χαίρομαι ιδιαίτερος ε, που ε, λαμβάνω εδώ το λόγο στην Επιτροπή σας, παραμονές της 25ης επαιτίου της υπογραφής της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Μάστριχτ. Εκείνη η τολμηρή απόφαση σηματοδότησε ε, μια νέα φάση στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και έθεσε τα θεμέλια της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Δέκα χρόνια μετά, οι πολίτες, οι Ευρωπαίοι πολίτες άρχισαν να έχουν χαρτονομίσματα ευρώ στα χέρια τους. Αυτό οδήγησε σε σημαντική ενίσχυση της πολιτικής δέσμευσης που μας κράτησε ενωμένους τα τελευταία 60 χρόνια. Είναι εύκολο να υποτιμήσει κανείς την ισχύ αυτής της δέσμευσης και της υπόσχεσης. Αλλά κάτι τέτοιο θα παρέβλεπε την ε, πρόοδο που έχουμε συντελέσει. Με το ενιαίο νόμισμα έχουμε σφυριλατήσει δεσμούς που άντεξαν τη χειρότερη οικονομική κρίση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και αυτό ουσιαστικά ήταν ο πραγματικός λόγος ύπαρξης του ευρωπαϊκού σχεδίου. Το να μας κρατήσει δηλαδή ενωμένους σε χαλεπούς καιρούς. Όταν ε, αναδύεται ο πειρασμός να στραφούμε κατά των γειτόνων μας ή να αναζητήσουμε εθνικές λύσεις. Ο στόχος όμως της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης θα έπρεπε να είναι να επιδιώξει την οικονομική και κοινωνική πρόοδο όπως ήταν και οι αρχικές προθέσεις ε, των μερών ε, της συνθήκης του Μάστριχτ. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε σταθερή ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Η ανθεκτική ανάκαμψη που διαπιστώσαμε και παρατηρήσαμε τον τελευταίο καιρό ήταν ένα ευπρόσδεκτο βήμα προς την υλοποίηση αυτού του στόχου. Την τελευταία διετία το κατακεφαλήν ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 3% στην Ευρωζώνη Κάτι που μας φέρνει σε καλή θέση σε σχέση με άλλες προηγμένες οικονομίες. Ε, η αίσθηση της οικονομικής κατάστασης ε, είναι καλύτερη, στο καλύτερο επίπεδο της τελευταίας πενταετίας. Η ανεργία έχει μειωθεί στο 9,6%. Το χαμηλότερο δηλαδή επίπεδο από το Μάιο του 2009. Και ο λόγος δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ μειώνεται για δεύτερη συνεχή χρονιά. Αυτά λοιπόν είναι βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση. Αλλά είναι μόνο τα πρώτα βήματα. Θα πρέπει να συνεχίσουμε σε αυτό το δρόμο, σε αυτή την άγουσα, ώστε να μειωθεί περαιτέρω η ανεργία, ώστε περισσότεροι Ευρωπαίοι να υποφεληθούν από την ανάκαμψη. Θα ξεκινήσω λοιπόν εξετάζοντας τη δική μας συνεισφορά για τη στήριξη της ανάκαμψης και θα σας εξηγήσω γιατί οι νομισματικές αποφάσεις του Δεκεμβρίου ήταν οι κατάλληλες και σωστές στο ισχύον οικονομικό πλαίσιο. Όπως μου ζητήσατε, θα αναφερθώ και στους κινδύνους στη χρηματοοικονομική χρηματοπιστική σταθερότητα που συνεχώς βρίσκονται υπό εποπτεία και παρακολούθηση. Η νομισματική μας πολιτική συνέβαλε τα μάλα στις ε, θετικές οικονομικές εξελίξεις που σας περιέγραψα πριν από λίγο. Τα μέτρα μας ε, ε, ωφέλησαν το χρηματοπιστωτικό σύστημα αλλά και την πραγματική οικονομία εξασφαλίζοντας πολύ ευνοϊκές χρηματοοικονομικές συνθήκες. Στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ ε, εντόπισε την ανάγκη της, ε, της μεγαλύτερης ενίσχυσης της ανάκαμψης προκειμένου να εξασφαλίσουμε υλοποίηση του στόχου της, του πληθωρισμού λίγο χαμηλότερα αλλά κοντά στο 2% μεσοπρόθεσμα. Και για να συμβεί κάτι τέτοιο θα πρέπει οι οικονομικές συνθήκες να μας υποστηρίζουν να είναι ευνοϊκές και λαμβάνοντας υπόψη τις αβεβαιότητες εντός και εκτός της Ευρωζώνης. Θα πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε τη συνέχιση της ποσοτικής χαλάρωσης και στο μέλλον. Με αυτό λοιπόν το υπόβαθρο αποφασίσαμε να παρατείνουμε το πρόγραμμα αγοράς περιουσιακών στοιχείων και πέραν του Μαρτίου του 2017 με πρόθεση να συνεχίσουμε τις αγορές μας μέχρι τα τέλη του Δεκεμβρίου του 2017 ή και ε, περαιτέρω αν παραστεί ανάγκη και εν πάση περιπτώσει μέχρι ότου το Διοικητικό Συμβούλιο δει πραγματική ε, πρόοδο στο στόχο υλοποίησης ε, του πληθωρισμού γύρω στα 2%. Θα συνεχίσουμε λοιπόν, ε, λοιπόν τις ε, αγορές μας σε ε, μηνιαίο επίπεδο 80 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το Μάρτιο και από τον Απρίλιο και μετά οι καθαρές μας αγορές θα είναι 60 δισεκατομμύρια το μήνα ενώ θα επανεπενδύσουμε τους τίτλους που έχουμε αγοράσει νωρίτερα στα πρόγραμμά μας στο μέτρο που πλησιάζουν προς τη λήξη τους. Αυτό θα ενισχύσει τις καθαρές μηνιαίες αγορές μας. Οι αποφάσεις του Δεκεμβρίου βρίσκουν τη σωστή ισορροπία μεταξύ της αυξανόμενης μας εμπιστοσύνης ότι οι οικονομικές προοπτικές Ευρωζώνης ενισχύονται και παγιώνονται και ταυτόχρονα δεν έχουμε σαφείς ενδείξεις σταθερής σύγκλησης των ποσοστών πληθωρισμού προς το επιθυμητό επίπεδο. Από τη μία πλευρά τα στοιχεία μας δείχνουν ότι ο ξύς κίνδυνος από πληθωρισμού έχει εκλείψει. Και ο πληθωρισμός ε, φαίνεται ότι θα αυξηθεί στο μέλλον. Αντίθετα προς την γενική αντίληψη, οι οικονομικές ε, συνθήκες ε, της Ευρωζώνης βελτιώθηκαν σταθερά. Η ανάπτυξη του ΑΕΠ στην Ευρωζώνη ήταν σταθερή κάθε τρίμηνο από την έναρξη του 2015, με μέσο όρο 1,9% το χρόνο. Σε σύγκριση με το 2013 έχουμε 3,5 εκατομμύρια λιγότερους ανέργους στην Ευρωζώνη. Μία μείωση δηλαδή άνω του 18%. Και το τελευταίο τρίμηνο η ανάκαμψη έχει επεκταθεί και σε άλλους κλάδους και σε άλλες χώρες. Και όντως αυτή η διαφορά του, της ανάπτυξης προστιθέμενης αξίας στις χώρες και τους κλάδους της Ευρωζώνης, αυτή η διαφορά έχει μειωθεί αισθητά και είναι σχεδόν ε, στα χαμηλότερα επίπεδα από την εισαγωγή του ενιαίου νομίσματος. Αλλά εξακολουθεί να είναι απαραίτητη η στήριξη από τα μέτρα νομισματικής μας πολιτικής αν θέλουμε πραγματικά τα ποσοστά πληθωρισμού να συγκλίνουν προς το στόχο μας με σταθερό και πάγιο τρόπο. Η αύξηση του ονομαστικού πληθωρισμού το Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο αντιστοιχεί σε σημαντικές ανωδικές συνέπειες όσο αφορά τη βάση και τις πρόσφατες αυξήσεις στις τιμές των ενεργειακών προϊόντων. Αντίθετα, οι πιέσεις του βασικού πληθωρισμού είναι ήπιες και μόνο σταδιακά θα αρχίσουν να αυξάνονται όσο προχωράμε. Αυτή η έλλειψη της όθησης όμως ό,τι αφορά τον υφέρποντα, το βασικό πληθωρισμό, αντικατοπτρίζει σε μεγάλο βαθμό τις πιέσεις ε, της ε, χαμηλής ε, εσωτερικής, του χαμηλού εσωτερικού εγχώριου κόστους. Και αυτό, δημιουργεί, και αυτό ε, οφείλεται και στην καθοδική πίεση σε ό,τι αφορά τους μισθούς λόγω της νοθρότητας αγοράς και της χαμηλής παραγωγικότητας. Όπως είπα και προηγουμένως, η νομισματική μας στρατηγική μας αναγκάζει να μην αντιδρούμε σε μεμονωμένα στοιχεία και σε βραχυπρόθεσμες αυξήσεις του πληθωρισμού ένας κατάλληλος ορίζοντας πολιτικής για μας είναι ο μέσο πρόθεσμος ορίζοντας. Γι' αυτό συνεχίζουμε να εξετάζουμε τις αλλαγές στον ενορμονισμένο δίκτυο τιμών καταναλωτή ε, και τις εξετάζουμε αν θεωρούμε ότι δεν ε, επηρεάζουν ε, σημαντικά την, το μέσο πρόθεσμο μας στόχο για σταθερότητα των τιμών. Επίσης, οι κίνδυνοι στις προοπτικές ευρωζώνης είναι χαμηλοί και σχετίζονται περισσότερο με παγκόσμιους παράγοντες. Η ισχύουσα νομισματική μας πολιτική και ο προσανατολισμός μας στην νομισματική πολιτική προβλέπουν ότι αν γίνει λιγότερο ευνοϊκός ο πληθωρισμός ή αν ε, οι χρηματοοικονομικές συνθήκες γίνουν ασύμβατες με περαιτέρω πρόοδο σε μια προσαρμογή του πληθωρισμού, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι έτοιμο να αυξήσει το πρόγραμμα αγοράς περιουσιακών στοιχείων και ως προς το μέγεθο και ως προς τη διάρκεια του. Μου ζητήσατε επίσης ε, να σχολιάσω και τις, ε, το πώς η διευκολυντική αυτή νομισματική μας πολιτική επηρεάζει τη χρηματοοικονομική σταθερότητα. Πιστεύω ότι τα προτερήματα της ε, πολιτικής μας υπερβαίνουν τα μειονεκτήματα και τις παρενέργειές της. Οι παρενέργειες και τα αρνητικά αποτελέσματα θα αντιμετωπιστούν κυρίως και εν ανάγκη από άλλες πολιτικές. Όπως είπα, η νομισματική μας πολιτική συνέβαλε τα μάλα ε, στη στήριξη της ανάκαμψης. Και μάλιστα τα μέτρα μας διαδραμάτισαν κέριο ρόλο στην διαφύλαξη της σταθερότητας της Ευρωζώνης, συμπεριλαμβανομένης και της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Θα ήθελα τώρα να πω λίγα λόγια για τις πιθανές παρενέργειες μιας υπερβολικά διευκολυντικής νομισματικής πολιτικής στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Μία από τις παράπλευρες αυτές ενέργειες είναι ο αντίκτυπος στην κερδοφορία των τραπεζών. Ας δούμε όμως κάποια στοιχεία. Μετά μια επιβράδυνση στην κερδοφορία στο πρώτο τρίμηνο του 2016, η κερδοφορία των τραπεζών της Ευρωζώνης ε, σταθεροποιήθηκε στο δεύτερο τρίμηνο με βάση κάποια προκατακτικά στοιχεία, οι εξελίξεις για το τρίτο τρίμηνο φαίνεται να ευθυγραμμίζονται με αυτές του δεύτερου τριμήνου. Η νομισματική πολιτική μπορεί να έχει αντίκτυπο στην κερδοφορία των τραπεζών με, πολλές, με πολλούς τρόπους και από πολλούς διάβλους. Η εκτίμησή μας είναι ότι ε, μέχρι στιγμής αυτά τα αποτελέσματα αλληλοεξοδετερώνονται Οι χαμηλές και αρνητικές, ε, τα χαμηλά και αρνητικά ποσοστά μπορούν να μειώσουν τα περιθώρια, καθαρά περιθώρια κέρδους, αλλά ταυτόχρονα στηρίζοντας την ανάπτυξη και την ανάκαμψη μάλλον, μια διευκολυντική τέτοια νομισματική πολιτική περιορίζει ε, τις ε, πιθανότητες χρεοκοπίας και τις, ε, τα αδικήματα. Και επίσης βελτιώνει την κατάσταση της ε, πίστης και των δανείων των οικοκυριών και των ε, επιχειρήσεων. Και αυτό είναι πολύ θετικό και για τις τράπεζες. Αυτό ήταν σημαντικό λοιπόν και στήριξε τα εισοδήματα των τραπεζών τον τελευταίο χρόνο. Επιπλέον, ε, χαμηλά μακροπρόθεσμα επιτόκια αυξάνουν, την αγοραία αξία των οικονομικών τίτλων που κατέχουν οι τράπεζες και αυτό οδηγεί σε κέρδη του κεφαλαίου που στηρίζουν περαιτέρω την κερδοφορία των τραπεζών. Και αυτή η συνολική εικόνα καλύπτει βέβαια κάποια ετερογένεια, ανομιομορφία που επικρατεί στον τραπεζικό τομέα. Και ιδιαίτερα ανάλογα με το επιχειρησιακό μοντέλο, επιχειρηματικό τους μοντέλο, οι μεμονωμένες τράπεζες μπορεί να επηρεαστούν με διαφορετικό τρόπο από ένα περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων. Ένα δεύτερο θέμα είναι ο δυνητικός κίνδυνος φούσκας των δανείων ή φούσκας των περιουσιακών στοιχείων των τίτλων. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε διάσει κριτήρια για τέτοια υπερτίμηση των τιμών των τίτλων. Και οι, τιμές και οι διαφορές στα ε, τα ομόλογα των επιχειρήσεων και οι τιμές των μετοχών είναι σε κανονικούς ε, ρυθμούς και οι τιμές ε, των ακινήτων είναι, αυξάνονται με μέτριο τρόπο. Παρόλο που υπάρχει ανομοιομορφία και πάλι μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης. Και μάλιστα αυτή την εκτίμηση στηρίζει το γεγονός ότι η αύξηση του δανεισμού είναι μέτρια. Κάτι που δείχνει ότι η αύξηση των τιμών των περιουσιακών στοιχείων δεν αυξάνει και την μόχλευση. Οπότε όσο περισσότερο ισχύσει αυτή η διευκολυντική πολιτική, τόσο μεγαλώνει ο κίνδυνος για ανεπιθύμητα αποτελέσματα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Για παράδειγμα, οι τιμές των στοιχείων του ενεργητικού μπορεί να αυξηθούν σε επίπεδα που δεν ευθυγραμμίζονται με τα θεμελιώδη στοιχεία, γιατί ίσως οι επενδυτές μπουν στον κίνδυνο να αναλάβουν περισσότερο κίνδυνο όταν οι αποδόσεις είναι χαμηλές. Τέτοιου είδους εξελίξεις ε, αντιμετωπίζονται περισσότερο με μακρο- και μικροπροληπτικά μέτρα και στρατηγική. Και ενώ η ενιαία μας νομισματική πολιτική στόχο έχει τη νομισματική σταθερότητα στην Ευρωζώνη στο σύνολό της, η μακροπροληπτική πολιτική και τα σχετικά μέτρα μπορεί να αντιμετωπίσουν τη, τους κινδύνους χρηματοπιστωτικής που ίσως δημιουργηθούν σε μερικά τμήματα των αγορών σε μεμονωμένες δικαιοδοσίες ή σε μεμονωμένες χώρες. Η αντιμετώπιση αυτών των δυνητικών κινδύνων στην πηγή τους θα μειώσει το κίνδυνο της μετάδοσης αυτών των κινδύνων και στην υπόλοιπη Ευρωζώνη. Οι μικροπροληπτικές πολιτικές βοηθούν επίσης στον περιορισμό της στρωτότητας των τραπεζών Γι' αυτό χαιρετίζω και τι προτάσει για τη μείωση του κινδύνου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που πευλήθηκαν τον περασμένο Νοέμβριο και που αναπτύσσουν περαιτέρω το νομικό πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ε, και θα συμβάλλουν στην αύξηση τη αντοχή και τη ανθεκτικότητα των τραπεζών. Εν κατακλείδη, όπω είπα και την περασμένη εβδομάδα στη Λιουμπλιάνα και όπω μα έχει δείξει και η κρίση, τα ωφέλη του ενιαίου νομίσματο μπορούν ε, να γίνουν πλήρως κατανοητά και να αξιοποιηθούν πλήρως όσο έχουμε πολιτικές και θεσμικά όργανα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο που θα εξασφαλίζουν τα ωφέλη τους για τους πάντες. Και όταν ε, ξεκινούσαμε την εισαγωγή του ευρώ, αναλάβαμε τη δέσμευση να ε, ακολουθήσουμε την άγουσα της θεσμικής και οικονομικής σύγκλησης. Η κρίση μας έχει δείξει ότι δεν θα πρέπει να χαλαρώσουμε αυτή τη δέσμευση γιατί εξακολουθεί και σήμερα να έχει σημασία στο μέτρο που θέλουμε να ενισχύσουμε την Οικονομική και Νομισματική Ένωση και την Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στις ισχύουσες αβεβαιότητες και προετοιμάζοντάς την για τις μελλοντικές προκλήσεις. Η αθεκτικότητα της Ευρωζώνης το 2016 παρά μια σειρά αρνητικών κραδασμών μας έδειξε ότι βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο Επίσης δείχνει ότι οι μεταρρυθμίσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο απέφεραν καρπούς ό,τι αφορά την οικονομική ανάπτυξη. Και στο μέτρο που βελτιώνεται η οικονομική κατάσταση και παρόλο που υπάρχουν προκλήσεις σε άλλες πολιτικές ε, που φυσικά μας τράβηξαν την προσοχή, δεν θα πρέπει να χαλαρώσουμε τις προσπάθειές μας ε, προκειμένου να καταστήσουμε την Οικονομική και Νομισματική Ένωση πιο ανθεκτική και με μεγαλύτερη ευημερία. Επίσης θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις αναπομείνωσες και γνωστές α, ε, τροτές, ε, τροτά χαρακτηριστικά σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Και γι' αυτό προσβλέπω στην συνεχή υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σε αυτό το δεύτερο μεσό της κοινοβουλευτικής θητείας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή και είμαι στη διάθεσή σας ε, για να απαντήσω σε ερωτήσεις. Thank Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχετε βεβαίω την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτούς τους φιλόδοξους και απαραίτητους στόχους. Δύο λεπτά σας υπενθυμίζω έχουμε για κάθε ερώτηση και πέντε συνολικά με πρώτο τον κύριο Μάιερ, Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και καλώς ήρθατε κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου και πάλι να σας συγχαρώ για τη δουλειά σας και να εκφράσω την υποστήριξή μας. Η κατάσταση με τα πραγματικά επιτόκια βλέπουμε ότι δεν έχει ε, φτάσει στο μηδέν ο ε, δεν είναι στο στόχο, είναι κάπου στα μισά του στόχου, μπορεί να ανέβει λίγο, ωστόσο πέφτουν τα επιτόκια, γιατί τα ονομαστικά επιτόκια παραμένουν σταθερά. Επομένως, νομισματική πολιτική ε, δίνει περισσότερη όθηση στην πραγματική οικονομία, σε μια στιγμή που, όπως είπατε και εσείς, η οικονομία παρουσιάζει καλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Επομένως, θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς θα θέλατε να δείτε την εξέλιξη των πραγματικών επιτοκίων ε, για τα επόμενα τρίμηνα. Η δεύτερη ερώτηση, περισσότερο μακροοικονομικού χαρακτήρα, στον κόσμο που ζούμε σήμερα δυστυχώς ε, διαγνώσκουμε κάποια σημάδια ότι η οικονομική παγκόσμια διαχείριση μπορεί να περάσει από μια πιο φιλελεύθερη ε, διαχείριση και διακυβέρνηση που υποστηρίζει περισσότερο το εμπόριο προς μια πιο προστατευτική, τουλάχιστον από πλευράς ορισμένων μεγάλων κρατών. Τι κίνδυνο μπορεί αυτό να σημάνει για την ευρωπαϊκή οικονομία και πώς θα τα αντιμετωπίζατε, πώς θα απαντούσατε σε, μια τέτοια, σε ένα τέτοιο κίνδυνο. Ευχαριστώ. Λέει ο κύριος Δράγκη. Κοιτάξτε. Οι όροι που προσδιορίσε το Διοικητικό Συμβούλιο για τους στόχους του πληθωρισμού είναι βασικά τέσσερις στον αριθμό. Ο πρώτος είναι ότι πρέπει να υπάρξει σύγκληση προς τον στόχο του πληθωρισμού κοντά αλλά κάτω από το 2% μέσω πρόθεσμα ή εν πάση περιπτώσει μέσα στον ορίζοντα της σχετικής οικονομικής πολιτικής. Δεύτερον, αυτή η σύγκληση πρέπει να είναι διαρκή, σταθερή, βιώσιμη. Δηλαδή δεν θέλουμε εξελίξεις ή πληθωρισμό που θα θεωρούνταν ή θα θεωρούσαμε μεταβατικό ή μεταβατικές. Τρίτος όρος πρέπει να είναι αυτόνομος ο πληθωρισμός, αυτοϋποστηριζόμενος. Και γιατί. Γιατί το τωρινές προβολές του προσωπικού μας για τον πληθωρισμό που προβλέπουν ένα ποσοστό πληθωρισμού σχετικά κοντά στους στόχους, δηλαδή κοντά αλλά κάτω από το 2% έως το 2019. Αυτές οι προβλέψεις λοιπόν λένε ότι το τωρινό επίπεδο της επέκτασης των χρηματοοικονομικών όρων θα διατηρηθεί. Άρα, οι προσδοκίες της αγοράς προδικάζουν τη διατήρηση αυτών των οικονομικών μέτρων. Τέταρτο στοιχείο, ότι ο στόχος που δεν πρέπει ποτέ να λησμονήσουμε είναι τα ποσοστά αυτά του πληθωρισμού να ισχύουν για ολόκληρη την Ευρωζώνη και τι μπορεί κάποιες χώρες να ε, παρουσιάζουν ποσοστά πληθωρισμού που μπορεί να παρουσιάζουν με ζωτικότητα προσέγγιση προς τον στόχο. Εμείς, και είναι η εντολή μας αυτή, έχουμε ως στόχο έναν πληθωρισμό που θα ισχύει για ολόκληρη την Ευρωζώνη. Θα ήθελα επίσης να προσθέσω ότι ο στόχος μας για τα ποσοστά του πληθωρισμού προσδιορίζεται και θα εξακολουθήσει να ε, προσδιορίζεται ως ονομαστικός πληθωρισμός. Βεβαίως θα πρέπει να ε, συνεχίσουμε και να υποστηρίζουμε έτσι ώστε τα, οι εξελίξεις για τον ονομαστικό πληθωρισμό να είναι ε, διαρκή σταθερές μεσοπρόθεσμες και για ολόκληρη την Ευρωζώνη. Επομένως, κοιτούμε και άλλες μορφές του πληθωρισμού, όπως άλλες ε, πιέσεις πληθωριστικές που ανέφερα και στην ε, εισαγωγική μου δηλώση. Η δεύτερη σας ερώτηση. Η απάντησή μου λοιπόν θα είναι, είναι λίγο νωρίς για να το κρίνουμε. Ακούμε με ανησυχία τις προστατευτικές ε, ανακοινώσεις προστατευτικών μέτρων, γιατί σε τελευταία ανάλυση η Ευρωπαϊκή Ένωση ολόκληρη έχει ε, θεσπιστεί, έχει θεμελιωθεί πάνω στο ελεύθερο εμπόριο, πάνω στις τέσσερις ελευθερίες. Και άρα όταν έρθει η ώρα και δούμε την εγκαθίδρυση των μέτρων που ανακοινώθηκαν, θα δούμε τι στάση θα τηρήσουμε. Ο κύριος Φολφαϊσέκερ από τους Σοσιαλιστές Δημοκράτες, Φον Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που σας βλέπω εδώ. Ήταν πιστικά τα επιχειρήματα που προβάλλατε στην εισαγωγική σας τοποθέτηση ότι η εντολή σας και τα μέτρα που αναπτύσσετε προχωρούν κατά τρόπο συντονισμένο, αντίθετα με αυτά που προβάλλουν ορισμένοι ε, επικριτές σε σχέση με τον ονομαστικό πληθωρισμό. Εξήγησε το βέβαια εσείς γιατί ο ονομαστικός πληθωρισμός σε ορισμένες χώρες να, μπορεί να μην είναι ο καλύτερος τρόπος για την ε, επίτευξη των στόχων και των, της εντολής σας. Ωστόσο είπατε κι εσείς ότι υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι συνδεδεμένοι με αυτή την πολιτική. Επομένως, ε, η ανθεκτικότητα και η αποδοτικότητα ορισμένων μέτρων θα κρίνουν την αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων. Και σας ρωτώ, Πώς νομίζετε ότι μπορούμε να το επιτύχουμε αυτό, δεδομένης της απόφασης του διατάγματος του Προέδρου Τραμπ που εκδόθηκε την Παρασκευή, σε σχέση με μέτρα τα οποία μπορεί να φαίνονται ότι είναι σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές ε, ρυθμίσεις, αλλά πάντως ρίχνουν στην πραγματικότητα διαφορετικό φως, δηλαδή βάζουν ένα αριθμό 120 ημερών, άρα σε τρεις φορές το χρόνο μπορεί να αποδιαρθρώνεται η πολιτική και όλα τα διδάγματα που έχουμε αποκομίσει από τις αγορές. Επομένως, θέλω να ρωτήσω, δεδομένων ε, δεδομένων των, της, δεδομένης της σημασίας, ε, της ευρωστίας και της, ε, του σχεδιασμού των μέτρων πώς μπορεί να απαντήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στις προκλήσεις αυτές. Και δεύτερον, πιο συγκεκριμένα, για κάτι που έχουμε αρχίσει να συζητούμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που είναι η η υπόθεση των κεντρικών αντισυμβαλωμένων ε, είναι το θέμα του γιατί έχουμε αποφασίσει να δημιουργήσουμε μια ε, τραπεζική ένωση και ως εκ τούτου ερωτώ πώς μπορείτε να Θεωρείτε ότι είναι ακόμη η καταλληλότερη προσέγγιση αυτή του ε, συλλογικού οργάνου των ρυθμιστικών αρχών εν ώψη των κεντρικών αντισυμβαλωμένων, που είναι πολύ μεγάλε τράπεζε ουσιαστικά. Απάντηση. Κοιτάξτε, για την πρώτη ερώτηση, θα έλεγα ότι σε ένα βαθμό είναι νωρί ακόμη για να βγάλουμε συμπεράσματα. Ωστόσο, αν δούμε τι μας διδάσκει η ιστορική εμπειρία, και, ποιοι, και διερωτηθούμε ποιοι είναι οι λόγοι και οι πηγές της χρηματοοικονομικής κρίσης που ξεκίνησε το 2007 και συνεχίστηκε μετά. Μπορεί κανείς να έχει διαφορετική εκτίμηση για το αν ήταν υπερβολικά επεκτατική η νομισματική πολιτική αυτός ο λόγος, η πηγή των προβλημάτων. Κάποιοι άλλοι μπορούν να λένε ότι πρόκειται για την αποδιάρθρωση των υφισταμένων ε, χρηματοοικονομικών ρυθμίσεων και κανόνων που είχε προηγηθεί. Αλλά νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουν πως πηγή των προβλημάτων του οικονομικών και της κρίσης ήταν ο συνδυασμός των δύο αυτών παραγόντων. Και αυτό το βλέπουμε ε, σε κάθε περίπτωση, σε κάθε ένα μεταξύ διαφορετικούς ε, ε, όρους ίσως ή βαθμίδες, αναλόγως και της εξέλιξης των διαφορών οικονομιών. Ως εκ τούτου, αυτό που δεν χρειαζόμαστε καθόλου αυτή τη στιγμή θα ήταν η χαλάρωση η ρυθμιστική των αγορών. Και σε μεγάλο βαθμό το γεγονός ότι δεν βλέπουμε εξέλιξη στους, σημαντικούς χρηματοοικονομικούς κινδύνους, αποτελεί και την ανταμοιβή της δράσης των ρυθμιστικών αρχών, των εποπτικών αρχών, για ό,τι έχουν κάνει από την ε, έναρξη της χρηματοοικονομικής κρίσης. Οι χρηματοπιστωτικοί διαμεσολαβητές αυτή τη στιγμή είναι πολύ πιο ισχυρή από ό,τι στην αρχή τη χρηματοοικονομική κρίση. Άρα λοιπόν δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει να επανέλθουμε στι ίδιε συνθήκε που είχαμε στην εκκίνηση τη ε, κρίση. Κάτι τέτοιο θα ήταν πάρα πολύ ανησυχητικό. Ελπίζω να απάντησα στην ερώτησή σα. Και για τη δεύτερη ερώτηση. για τους CCPs για τους κεντρικούς αντισυμβαλόμενους. Υπάρχει μια πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εμείς υποστηρίζουμε την ενίσχυση των ρυθμίσεων για την εξυγίαση των κεντρικών αντισυμβαλωμένων μέσα σε ένα πλαίσιο το οποίο πρέπει να επανεξεταστεί. Πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρέπει να διαδραματίσει ρόλο στη ρύθμιση των κεντρικών αντισυμβαλωμένων και Εν τέλει, η αδίποτε ρύθμιση πρέπει να είναι σύμφωνη με τις διεθνείς προδιαγραφές και τα πρότυπα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μαριάς, παρακαλώ, ECR. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Ντράγκη, η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στη διαδικασία αναδιάρθρωσης του ελληνικού δημοσίου χρέους, το γνωστό PSI, που έγινε το 2012 στην Ελλάδα, οδήγησε στο κούρεμα κατά 53,5% των ομολόγων των ιδιωτών, των μικροομολογιούχων φυσικών προσώπων. Πάνω από 15.000 μικρομολογιούχοι λοιπόν έχασαν πάνω από 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Έναντι του υπολείπου 46,5% του κεφαλαίου τους, το 31,5% αντικαταστάθηκε από ομόλογα του ελληνικού δημοσίου τα οποία ξεκινούν από το 2023 μέχρι το 2042 να πληρώνονται. Έτσι, σε αντίθεση με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία απέφυγε το κούρεμα στο PSI και γλίτωσε 54 δισεκατομμύρια ευρώ, οι μικροομολογιούχοι φυσικά πρόσωπα, εάν εξοφληθούν ποτέ, θα μπορέσουν να εξοφληθούν το 2042, εάν ζουν βέβαια μέχρι τότε προκειμένου να θεραπευτεί αυτή η αδικία, θα ήθελα να σας υποβάλω μία πρόταση και να μου απαντήσετε. Εάν το ευρωσύστημα και ειδικότερα η ΕΚΟΥΤΟΥ και η Τράπεζα της Ελλάδος, στο πλαίσιο του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης, θα μπορούσαν να προχωρήσουν εντός του 2017 στην αγορά των ομολόγων αυτών του ελληνικού δημοσίου, καταβάλλοντας τα ποσά στους δικαιούχους και εξοφλώντας τους στο 100% όλα τα ομόλογα που λήγουν από το 2022 μέχρι το 2042. Με αυτόν τον τρόπο η ΕΚΤ θα συμβάλλει στην αποκατάσταση μιας αδικίας, το κόστος είναι περίπου 800 εκατομμύρια ευρώ και έτσι θα έχουμε τη δυνατότητα η ΕΚΤ να δράσει επιτέλους για ποσοτική χαλάρωση υπέρ των πολιτών, δηλαδή το γνωστό QE for People. Θα ήθελα μια απάντηση στο θέμα αυτό κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την πρώτη σας ερώτηση. Το μόνο που μπορώ να πω σε αυτό το στάδιο είναι ότι οι όροι της αναδιάρθρωσης προσδιορίστηκαν την εποχή εκείνη και εξ όσων γνωρίζω εγώ δεν υπάρχει πρόθεση αναθεώρησης των όρων της αναδιάρθρωσης. Αν όμως ε, έχω τη δυνατότητα για μια πληρέστερη απάντηση, πολύ ευχαριστώ να σας τη στείλω γραπτός. Για το δεύτερο τμήμα, επιτρέψτε μου να επιμείνω γιατί είναι μια ερώτηση που μου επανέρχεται συνεχώς. Πότε θα αγοράσει και αν θα αγοράσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τραπέζα ελληνικό χρέος. Πρώτον πρέπει να δούμε πρώτα απ' όλα, πρώτα απ' όλα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της βιωσιμότητας του χρέους. Για να φτάσουμε σε μια πιστική αξιολόγηση της βιωσιμότητας του χρέους βράχη αλλά και μακροπρόθεσμα μέτρα, πρόθεσμα ήδη έχουν τεθεί σε εφαρμογή, αλλά και τα, τα τα οποία βρίσκονται από διαπραγμάτευση μεταξύ των κρατών μελών, πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή. Έτσι μπορεί να γίνει μια πιστική αξιολόγηση της βιωσιμότητας του χρέους. Με άλλα λόγια, πρέπει να ολοκληρωθεί η, η αξιολόγηση, η δεύτερη αξιολόγηση. Άπαξ και συμβεί αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόλυτη ανεξαρτησία θα εκφράσει τη δική του αξιολόγηση αυτής της βιωσιμότητας με βάση και μελήματα αξιολόγησης, διαχείρισης καλύτερα κινδύνου. Και τότε μόνο μπορούμε να μιλούμε για αγορά χρέους. Μπορεί να βρισκόμαστε κοντά στο στόχο αυτόν εάν έρθει η αξιολόγηση, η δεύτερη αξιολόγηση σχετικά σύντομα ή μπορεί να περάσει περισσότερο διάστημα χρονικό πριν φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση. Ε, είχα μερικά δευτερόλεπτα, Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να συνεχίσω. Κύριε Ντράγκη, η ερώτησή μου είναι πολύ συγκεκριμένη για τους μικρομολογιούχους οι οποίοι κατεστράφησαν. Εάν δηλαδή αποφασίσετε να αγοράσετε ελληνικό χρέος, θα μπορέσετε να προαγοράσετε τα ομόλογα των μικροομολογιούχων και να τους εξοφλήσετε στο 100% παρότι λήγουν το 2042. Θέλουν μια απάντηση. Σας παρακολουθούν χιλιάδες άνθρωποι. Το θέμα είναι σοβαρό. Ευχαριστώ. Ασφαλώς και θα εξετάσουμε αυτή την ιδέα, αλλά δεν πρέπει να λησμονούμε ότι οι κανόνες που διέπουν τις αγορές ισχύουν για όλες τις χώρες μέλη. Άρα πρέπει να ξεκινήσουμε από την ίδια βάση, από τις ίδιες αρχές και προδιαγραφές. Ευχαριστώ. Ελπίζουμε λοιπόν να ολοκληρωθεί ομαλά η δεύτερη αξιολόγηση. Από την Άλντε η κόρη Νόη Βαρχόλτσεν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. καλώ ήλθατε κύριε Ντράγκη. Δύο ερωτήσει. Η πρώτη αφορά την νομισματική πολιτική και η δεύτερη την κυβερνοασφάλεια. Είπατε και ο ίδιο ε, στην εισαγωγική σα παρέμβαση ότι η νομισματική πολιτική σας δεν θα σας κάνει και τον πλέον δημοφιλή στις χώρες, μεταξύ ε, και, της, και στη δική μου χώρα. Πρέπει να σας πω ότι θεωρούμε ότι παίρνετε πολλά νομισματικά στεροειδή για να τονώσετε την οικονομία Τέλος πάντων, είπατε επίσης ότι η νομισματική πολιτική δεν μπορεί να συνεχίζεται επαόριστον. Και επίσης αντιλαμβάνουμε ότι το σενάριο στρατηγική εξόδων. Θέλετε, δεν μπορείτε να τα συζητήσετε λεπτομεριακά μαζί μας. Επισκεφτήκατε όμω με αντιπροσωπεία ε, τη ΕΚΟΝ ε, τη ΕΠΑ και data-driven, μας είπε η ΦΕΔ ότι είναι η πολιτική, όχι date-driven, δηλαδή βασίζεται στα δεδομένα και όχι σε ημερομηνίε. Ε, το ίδιο σχέδιο για την πολιτική της ΕΚΤΑ και αν ναι, τι δεδομένα λαμβάνετε υπόψη σας, τι στοιχεία. Δεύτερη ερώτηση, ε, κυβερνοχώρος. Ε, Φραγκφούρτη το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Εκεί ε, αναφερθήκατε με πολύ θετικά λόγια στις δυνατότητες ε, των νέων τεχνολογιών για το χρηματοπιστωτικό τομέα, καινοτομία και επειδή είμαι για την FinTech, συμφωνώ με τα χαράς μάλιστα μαζί σας και πιστεύω ότι πράγματι θα πρέπει να έρθουν σε αίσιο πέρα όλα αυτά και οι νέε εξελίξει. Όμω υπάρχουν και οι απειλέ στον κυβερνοχώρο, οι κίνδυνοι ε, για την ασφάλεια. Πιστεύετε λοιπόν ότι η κυβερνοασφάλεια στο χρηματοπιστωτικό τομέα είναι αρκετά ψηλά στον κατάλογο προτεραιοτήτων, στι δοκιμέ κόπου αντοχή, στα λεγόμενα stress test, ή μήπω πρέπει να αναβαθμιστούν. Γνωρίζουμε αρκετά, έχουμε αρκετή εμπειρία ε, στο επίπεδο των εποπτικών αρχών ή θεωρείτε ότι χρειάζεται κάτι παραπάνω. Ευχαριστώ απάντηση. Να απαντήσω στο δεύτερο καταρχάς ερώτημα. Φυσικά και πρέπει να αναβαθμίσουμε τις προσπάθειες η εμπειρία μας με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο τα τελευταία 4-5 χρόνια μας δείχνει ότι πολλές φορές ε, πιαστήκαμε προετοίμαστοι, όχι μόνο στο χρηματοπιστωτικό τομέα, αλλά γενικότερα. Επομένως, υπάρχει ένα σοβαρό, θα, για να μην πω κβαντικό άλμα, ένα ποιοτικό άλμα που πρέπει να γίνει από όλους και από τις χρηματοπιστωτικές ε, υπηρεσίε και μιλώ και για τον ιδιωτικό ε, κλάδο, τους, τις αποτικές αρχές επίσης, που πρέπει να κάνουν αυτό το ποιοτικό άλμα. Και σε ό,τι αφορά τα ε, benchmarks, αυτά τα μέτρα σύγκρισης, ξέρετε, οι κυβερνοαπειλές εξελίσσονται, μεταβάλλονται και με την τεχνολογία και την καινοτομία επίσης. Επομένως, σίγουρα ε, επειδή δεν είναι πεπερασμένο αυτό το πρόβλημα, θα πρέπει να συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε πιο ασφαλή και καλύτερα πρότυπα και κανόνες. Και έρχομαι στο πρώτο σας ερώτημα τώρα. Τι χρειάζεται για να γίνει σαφές ποιο θα είναι το επόμενο βήμα. Ουσιαστικά χρειάζεται ένας δείκτης ε, πληθωρισμού που θα πληρεί τέσσερις προϋποθέσεις, οποίες και προανέφερα. Δηλαδή σύγκληση προς τους στόχους, βιώσιμη σύγκληση, μεσοπρόθεσμα, δηλαδή, δηλαδή ε, σε έναν ορατό ορίζοντα. Επίσης θέλουμε μια αυτάρκη αν θέλετε, ε, αυτοσυντηρούμενη κατάσταση. Ας υποθέσουμε ότι δεν υπάρχει πλέον η δική μας στήριξη. Τι θα συμβεί. Θα υπάρξει αυτή διαμείωση του δίκτυου πληροφορισμού ή θα συνεχίσει τη σύγκληση προς του μεσοπρόθεσμου στόχους. Ε, και βέβαια η απάντηση είναι η δεύτερη. Αν ισχύει αυτή η προϋπόθεση λοιπόν, τότε μπορούμε να αποσύρουμε ε, την νομισματική στήριξη. Τέταρτη προϋπόθεση δεν θα κουραστώ και δεν θα σταματήσω ποτέ να το λέω σε όλες τις χώρες και στη δική σας, ότι δηλαδή η δίκτυση του πληθωρισμού θα πρέπει να αφορά όλη την Ευρωζώνη. Γιατί μόνο ε, έτσι ορίζεται άλλωστε και η δική μας εντολή κατά αυτόν τον τρόπο. Ευχαριστώ η Μαρίσα Ματίας από την ΚΟΕ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και εσάς κύριε Ντράγκη. Η Ευρωζώνη το 2016 ε, τελείωσε με κάτω από το 2% και ε, τον Ιανουάριο του 2017 αυξήθηκε ο πληθωρισμός μεν, αλλά όχι σε όλα τα προϊόντα και από το 2012 η ΕΚΤ παραβιάζει συστηματικά την εντολή της. Και παρά τις δυσκολίες αυτές και παρά τις παραβιάσεις εντολής, το θέμα της ποσοτικής χαλάρωσης είχε πολύ μέτρια αποτελέσματα για την οικονομία και για την ε, ανάκαμψη στα κράτη-μέλη. Και μάλιστα, ενώ ε, δεν ε, υλοποιούμε το στόχο του πληθυσμού, αυξάνουμε τα ενάψματα. Αυτό οδήγησε σε αύξηση του δημόσιου χρέους της Πορτογαλίας, παρόλο που η Πορτογαλία ευνηδίασε όλες τις, όλα τα κοινωτικά θεσμικά όργανα και ε, κατάφερε να μειώσει το έλλειμμα της. Επίσης, πώς γίνεται η κατανομή στο πρόγραμμα αγορών του ΕΚΤ. Γιατί εξαιτία ε, του υψηλού δίκτυου ε, χρέου που έχει η Πορτογαλία δεν έχει πρόσβαση στι αγορέ από την ΕΚΤ, παρόλο που τι δικαιούται. Αυτό είναι μια παράδοξη εξωφρενική κατάσταση. Γιατί έχουμε τον ίδιο λόγο χρέου ΑΕΠ με την Ιταλία. Έχουμε υψηλότερο πρωτογενέ πλεόνασμα, αλλά καταβάλουμε στην Πορτογαλία ψηλότερα επιτόκια γιατί δεν έχουμε πρόσβαση στο πρόγραμμα αγορών της ΕΚΤ. Σε αντίθεση με την Ιταλία που έχει υπερβεί το, την κλίδα κεφαλαίου, ενώ εμείς δεν έχουμε φτάσει ακόμη στην κλίδα κεφαλαίου. Γι' αυτό έχω κάποιες απλούστατες ερωτήσεις. Καταρχήν, ως προς την ιδέα της ισοτιμίας, της ισότητας μεταξύ των κρατών μελών. Είπατε ότι συμμερίζετε αυτήν την ιδέα ότι όλες οι, όλες οι χώρες είναι ισότιμες. Θα προβλέψετε λοιπόν κάποιο μηχανισμό αντιστάθμισης, μια και ε, στην πράξη δεν έχουμε σήμερα ισότητα μεταξύ των κρατών μελών και μάλιστα επιδεινώνεται η κατάσταση και θα επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο το 2017. Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρόκειται να επανεπιταχύνει το πρόγραμμα της ποσοτικής χαλάρωσης ή θα το μειώσει ή θα συνεχίσετε να παραβιάζετε την εντολή για την οποία εκλεγήκατε, όπως κάνετε μέχρι στιγμής. Ευχαριστώ. Για το πρώτο σας ερώτημα, την επιτυχία δηλαδή της νομισματικής μας πολιτικής ε, Φυσικά και θα ε, μιλήσω μεροληπτικά, αλλά εγώ θεωρώ ναι ότι είναι επιτυχημένη η νομισματική πολιτική και το βλέπετε. Βλέπετε την επιτυχία σήμερα. Εκατομμύρια θέσεις εργασίας δημιουργούνται. Το είπα και στην εισαγωγική μου παρέμβαση. Αυτό είναι απόδειξη. Βαθμιδών η ανάκαμψη προχωρά, σταθερά. Έχουμε ανάπτυξη από τις αρχές ε, ε, του 2015, τρίμηνο το τρίμηνο, σταθερά. Θα δούμε όλα αυτά πώς θα μεταφραστούν σταδιακά ε, σε αύξηση των ονομαστικών μισθών και σε υψηλότερη ανάπτυξη των τιμών, όχι λόγω της ενέργειας, αλλά και των άλλων συστατικών του δίκτυ τιμών καταναλωτή. Ε, θεωρώ λοιπόν ότι ήταν επιτυχής μέχρι τώρα νομισματική μας πολιτική. Επίσης, αν εξετάσετε και τις χαμηλές τιμές πετρελαίου και λάβετε υπόψη σας και αυτό τον παράγοντα, έστω μέχρι πριν από λίγους μήνες, οι δύο μοχλοί της ανάκαμψης ήταν ακριβώς οι χαμηλές τιμές πετρελαίου και η δική μας νομισματική πολιτική. Δεν υπήρχε και τίποτε περισσότερο επί σειρά ετών ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη. Δεύτερο ε, τμήμα του πρώτου σας ερωτήματος. Μιλήσατε για τα spread, για το χρέος ε, των κρατών μελών. Η δική μας νομισματική πολιτική δεν στοχεύει στα spread, αλλά τη σταθερότητα των τιμών. Αυτός είναι ο στόχος της πολιτικής μας, όχι τα spread. Πάντα το πρώτο σας ερώτημα, ένα τρίτο κομμάτι είχε να κάνει με την υποτιθέμενη άνηση μεταχείριση μεταξύ χωρών. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει καμία άνηση μεταχείριση. Θα πρέπει να έχετε υπόψη ότι υπάρχουν και όρια σε ό,τι αφορά την έκδοση. Επομένως, το πρόγραμμα αγοράς περιουσιακών στοιχείων βλέπει και, ε, ε, και το θέμα αυτό. τις κλήθες κεφαλαίου αλλά και τα όρια στις εκδόσεις. Δεσμευόμαστε και το οικονομικό, ε, μάλλον το Διοικητικό Συμβουλίο το ανέφερε πρόσφατα λόγω αυτών των ορίων όπως σας είπα. Σε ό,τι αφορά τώρα, ναι το είπα και στην εισαγωγική μου παρέμβαση, αν οι όροι χρηματοδότησης δεν συνέπιπταν ε, με τις προσπάθειες εκπλήρωσης ε, του στόχου μας γύρω στο 2% ε, όπως είπα μέσω πρόγραμμα για όλη την Ευρωζώνη με βιώσιμο τρόπο, τότε ναι, θα επέμβουμε εκ νέου. Θα αυξήσουμε το πρόγραμμα αγοράς, θα το ενισχύσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Φίλιπ Λάμπερτς από τους Πρασίνους. Ευχαριστώ και καλησπέρα σας κύριε Πρόεδρε όταν σας ακούω να μιλάτε για απασχόληση και ανάπτυξη, αν θέλετε άπειρη ανάπτυξη σε ε, περασμένο κόσμο, θα πρέπει να αποσυνδέσετε την, την ανάκαμψη από, το, από την, τον υλικό παράγοντα, κάτι που δεν γίνεται, θα, το έλεγε αυτός ο μηχανικός. Αλλά το θέμα είναι ε, τι γίνεται με την απασχόληση, όχι την ανεργία. Είναι 68 στην ε, Γερμανία, 63 στο Βέλγιο, 65 στην Ιταλία, οπότε θα, θέλαμε πολύ μεγαλύτερη ανάπτυξη για να επιτύχουμε την πλήρη απασχόληση που είναι ο στόχος. Επίσης, ε, σε ό,τι αφορά το στόχο της ε, σταθερότητας των τιμών, και ο τρόπος που τερμινεύεται αυτό το άρθρο είναι γύρω ή κάτω από το 2%. Δεν υπάρχει άλλος ορισμός της ε, σταθερότητα των τιμών. Διαβάζοντα και πάλι το άρθρο 127, βλέπω ότι παραπέμπει στο άρθρο 3 τη συνθήκη, που αναφέρεται στην κοινωνική πρόοδο, στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα και ούτω καθεξής. Οπότε ρωτώ, ε, ποιος είναι ο τρόπο με τον οποίο κατανέμεται ο αντίκτυπο τη νομισματική πολιτική τη ΕΚΤ. Βέβαια υπάρχει το θέμα τη ποσοτικής χαλάρωση που μερικέ φορέ έχει αρνητικά αποτελέσματα, αλλά πώ. ε, επηρεάζει τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις ε, που στηρίζει η ΕΚΤ. Και εμείς θέλουμε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, αλλά διαφορετικές από αυτές που πρεσβεύετε εσείς. Σε ό,τι αφορά τη μόνιμη ε, ελαστικοποίηση της αγοράς εργασίας, αυτό έχει μια αρνητική πανέργεια στην κατανομή του εισοδήματος. Γιατί φαίνεται τους ε, εργαζόμενους ανταγωνισμό μεταξύ τους και έτσι επιτρέπεται στο κεφάλαιο να εξάγει μεγαλύτερη ε, προστιθέμενη αξία. Τι έχετε να απαντήσετε σε αυτά. Η απάντηση στην πρώτη ερώτηση είναι θετική, ότι για μας ο μόνος, ο μόνος σωστός ορισμός της ε, σταθερότητας των τιμών είναι αυτός που αφορά τον πληθωρισμό γύρω κάτω από το 2%. Κάτω από το 2% αλλά κοντά στο 2%. Και αυτό ε, μας καθοδηγεί στην νομισματική μας πολιτική. Δεύτερον, εξετάζουμε με ιδιαίτερη προσοχή τον αντίκτυπο που έχει στην κατανομή του εισοδήματος ε, η πολιτική μας της ποσοτικής χαλάρωσης. Πριν από λίγους μήνες ε, έκανα μία ομιλία στο Βερολίνο και εκεί με εξονυχιστικές λεπτομέρειες έκανα μία ανάλυση του διανεμητικών συνεπειών της νομισματικής μας πολιτικής. Πάντως θα μπορούσε κανείς γενικά να πει ότι η νομισματική μας πολιτική αντιμετωπίζει τις ε, κυριότερες συνέπειες ε, της ανισότητας ε, στις κοινωνίες μας, που είναι κυρίως η ανεργία. Και από αυτή την άποψη είχε μεσοπρόθεσμες συνέπειες η ποσοτική μας χαλάρωση, που μάλιστα περιόριζαν την ανισότητα. Βέβαια, είναι αλήθεια ότι βραχυπρόθεσμα όσο αγοράζουμε περιουσιακά στοιχεία και η τιμή τους αυξάνεται και φυσικά κάτοχος των ε, περιουσιακών στοιχείων δεν είναι, ε, δεν είναι τα φτωχότερα τμήματα του πληθυσμού. Οπότε βράχει πρόθεσμα ίσως το αποτέλεσμα διανεμητικά δεν θα ήταν πολύ θετικό. Αλλά δεν είναι και πολύ αρνητικό για πολλούς και διάφορους λόγους. Για παράδειγμα, έχουν αυξηθεί τιμές των ακινήτων των κατοικιών και η ιδιοκτησία όμως των κατοικιών είναι σχετικά δίκαια κατανεμημένη στην κοινωνία. Και τα μεσοπρόθεσμα αποτελέσματα της ποσοτικής χαλάρωσης σίγουρα είναι θετικά ως προς την ανισότητα. Σε ό,τι αφορά τι διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσει, κατά πάσα πιθανότητα ε, οι δικέ σα δεν ε, είναι απόλυτα συμβατέ με τις δικέ μου, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχουν και μεγάλε διαφορέ. Και τώρα, Σίγουρα κάθε χώρα έχει το δικό της πρόγραμμα για τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Σε μετρηπικές χώρες έχουμε θέματα όπως η δικαιοσύνη, η παιδεία. Σε άλλες χώρες οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις αφορούν την αγορά εργασίας. Πάντως σε όλες τις χώρες, και αυτό θα πρέπει να είναι το πρώτο ζητούμενο, είναι η ολοκλήρωση της ε, ενιαίας αγοράς. Δηλαδή, ο ανταγωνισμός και οι εμπορικές συναλλαγές, αγαθά και υπηρεσίες. Και όπω δείχνει και η μακροοικονομική θεωρία, αυτό πρέπει να είναι και ο πρώτο στόχο, η πρώτη διαρθρωτική μεταρρύθμιση που υλοποιείται. Βέβαια, έχουμε και άλλε που έπονται, αγορά εργασία, δικαιοσύνη, παιδεία, όπου χρειάζονται και αυτέ. Υπάρχει όμω και μία άλλη πτυχή με την οποία συμφωνώ και ίσως έχει παραβλεφθεί κάπως τελευταία χρόνια, Όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις προϋποθέτουν τεράστιες αλλαγές στις κοινωνίες μας. Και οι ρηξικέλευθες αλλαγές δημιουργούν νικητές και χαμένους. Και τους χαμένους θα πρέπει να τους προσέξουμε πολύ περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν. Και αν δείτε τα βασικά μας εγχειρίδια Πάντα λέγαμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα είδο αντιστάθμιση ή αποζημίωση σε περίπτωση που γίνονται ρηξικέλευτε αλλαγέ στην κοινωνία. Και υπάρχουν τρόποι να λάβουμε υπόψη και του χαμένου. Θα πρέπει λοιπόν και αυτό να, σκεφτούμε, να μην τους αγνοήσουμε δηλαδή. Σας ευχαριστώ. Ο Μάρκο Τζάνι από την ΕΝΕΦ. Πρόεδρε Τράκη, Έχετε ασφαλώ παρακολουθήσει τη συζήτηση που αναπτύχθηκε μεταξύ ΗΠΑ και Γερμανίας μετά τις κατηγορίες ε, του Πρόεδρου Τραμπ προς τη γερμανική κυβέρνηση ότι χειραγωγεί την ισοτιμία και η γερμανική κυβέρνηση είπε ότι υπεύθυνη ήταν η πολιτική, νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τις ανισότητες αυτές. Μάλιστα ότι, την είχε, ότι σας είχε προειδοποιήσει και ότι παρόλα αυτά προχωρήσατε προς αυτές τις επιλογές. Ερωτώ λοιπόν, εσείς συμφωνείτε με το Σόιμπλε ή νομίζετε ότι το πολύ χαμηλό επιτόκιο της Γερμανίας και ως εκ τούτου το εμπορικό της πλεόνασμα είναι κάτι το οποίο έχει προκύψει ύστερα από μια πολιτική εμονική για πλεονάσματα και κάτι άλλο, ύστερα από την ε, συζήτηση και την ομιλία που είχατε την προηγούμενη εβδομάδα στη Λουμπλιάνο, όπου επιτεθήκατε κατά των πολιτικών ορισμένων κρατών μελών, όπου είπατε τα κράτη που έχουν προβήσει σε μεταρρυθμίσει δεν έχουν ανάγκη από ευελιξία νομισματική για να εξασφαλίσουν μια σταθερότητα νομισματική. Μπορείτε λοιπόν κατόπιν αυτών των δηλώσεων να μα εξηγήσετε πώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μέσα από την εντολή τη έχει προβάλει νομισματικέ πολιτικέ οι οποίε υποτίμησαν το ευρώ κατά σημαντικό μάλιστα ποσοστό έναντι του ε, δολαρίου προκειμένου ε, να στηρίξουν την ανάπτυξη και μπορείτε να μας δώσετε κάποια παραδείγματα κρατών, μεγάλων κρατών της Ευρωζώνης που μπόρεσαν να υποφεληθούν από αυτή την ανάπτυξη και έχουν υψηλότερα ποσοστά ανάπτυξης του ΑΕΠ τους από τα μεγάλα κράτη πάντα της, Ευρωπαϊκής, της Ευρωζώνης από το 1999 μέχρι το 2015 με πολύ χαμηλότερα ε, επιτόκια από αυτά τα οποία χαρακτηρίζουν την οικονομία των ΗΠΑ και του ΗΠΑ και επίσης για την Ευρωζώνη. Πώς βλέπετε την επάνωδο σε μια δεύτερη εκδοχή της νομισματικής ε, ένωσης SME ε, με διακυμάνσεις μεταξύ των εθνικών νομισμάτων. Τι γλώσσα να μιλήσω, Πρόεδρε, για να απαντήσω. Ό,τι θέλετε. Για την πρώτη σας ερώτηση. Θα σας αναγνώσω ένα ενδιαφέρον έγγραφο. που πραγματεύεται το αν πράγματι εμείς χειραγωγούμε το νόμισμα ή όχι. Η τελευταία έκθεση προς το Κογκρέσο του Οκτωβρίου 2016 σε 14 Οκτωβρίου καταγράφει από πλευρά του ίδιου του US Treasury, του Υπουργείου των Οικονομικών, ότι δεν χειραγωγεί τη η Γερμανία και ο λόγο είναι ότι η Γερμανία δεν πληρεί τα τρία κριτήρια τα οποία ε, χρησιμοποιεί το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ για να εντοπίσει αθέμητε πολιτικέ επιλογέ και προγράμματα και ω εκ τούτου έχει σημαντικό ε, διμερές ε, πλεόνασμα μεν σε εμπορικούς όρους, αλλά δεν είναι αυτό σταθερό σε σχέση με μια παρέμβαση στην αγορά. Και συνεχίζουμε το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, το οποίο δηλώνει στην έκθεση πως διαπιστώνει πως δεν πληρεί ε, μία από τις οικονομίες που μελέτησε τα τρία αυτά κριτήρια. Η Γερμανία έχει και σημαντικό ε, διμερές πλεόνασμα και δεν έχει η ΕΚΤ παρεμβεί στις αγορές ε, των ισοτιμιών από το 2011 και κατόπιν μιας ε, σταθερής παρέμβασης ε, του G7 για τη σταθεροποίηση του ΓΕΝ σε συνεργασία με τις αρχές των ΗΠΑ και στα Ιταλικά, πρώτα απ' όλα δεν είμαστε χειραγωγή του νομίσματος. Δεύτερον, οι νομισματικές πολιτικές που ακολουθήσαμε αντικατοπτρίσουν, αντικατοπτρίσουν μια θέση αντιστάθμισης του κύκλου της Ευρωζώνης του, στις ΗΠΑ. Και ως εκ τούτου, το 2013, θα σας πενθυμίσω, ήταν 1,40 η ισοτιμία με το δολάριο. Το γερμανικό πλεόνασμα λοιπόν ήταν ήδη στο 6% σχέση με τις ΗΠΑ, το εμπορικό πλεόνασμα. Γιατί, γιατί αυτή είναι η δύναμη της γερμανικής οικονομίας που δεν στηρίζεται σε αυτό το οποίο εσείς χειριζόσαστε, δηλαδή την ε, καταχρηστική πολιτική στην αγορά εργασίας, αλλά και στην παραγωγικότητα και τον ανταγωνισμό που δεν στηρίζεται μόνο στις τιμές. Ποιες είναι οι χώρες που επωφελήθηκαν και που μπόρεσαν γιατί δεν θα συμφωνήσω καν ότι είχε λιγότερη ανάπτυξη ευρωζώνη σε σχέση με, άλλα, με άλλες περιοχές, φερειπίν ε, χώρες εκτός του ευρώ. Πολλές είναι χώρες που ανέφερα και τώρα στην ομιλία του, αλλά και στην ομιλία της Λουμπλιάνα, που πήγαν πολύ καλά παρά την κρίση. Πρώτη-πρώτη Γερμανία, αλλά και άλλες. Και η Ιρλανδία. Ακόμα και η Ιρλανδία. Δεν έχω τα στοιχεία μπροστά μου. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, και πάλι παρά την πολύ σοβαρή κρίση του ε, δημόσιο αλλά και του ιδιωτικού χρέους μπόρεσε να μειώσει την ανεργία η Ιρλανδία κατά πολύ σημαντικό ε, τρόπο. Οι κάτω χώρες, αλλά και πολλές άλλες χώρες που τα έχουν πάει καλά τα τελευταία χρόνια. Και το κατάφεραν σε μεγάλο βαθμό με, ε, χάρη στις διαρθωτικές τους μεταρρυθμίσεις που κατέστησαν πιο ισχυρές ε, τις οικονομίες τους, πιο ε, έτοιμες για ανάπτυξη. Στα αγγλικά. Και εν τέλει, για, μια δεύτερη, για ένα δεύτερο νομισματικό μηχανισμό που αναφέρατε SME2. Θα υπενθυμίσω τα λόγια του Προέδρου Ρέιγκαν σε μια προεκλογική εκστρατεία που είπε «Πάλι τα ίδια, μα σας παρακαλώ, είδαμε τι συνέβη με τις υπερβολικές ρυθμίσεις τις νομισματικές πριν από την εισαγωγή του ευρώ. Η δεκαετία του 70, η δεκαετία του 80 δεν χαρακτηριζόταν από σταθερότητα χαρακτηριζόταν διαρκώς από ανταγωνιστικές υποτιμήσεις νομισμάτων. Το όφελος θα ήταν ότι δεν θα είχε μπορέσει να επιβιώσει η εσωτερική αγορά, η ενιαία αγορά, με διαρκείς ανταγωνιστικές υποτιμήσεις νομισμάτων. Ευχαριστώ Μάρκο Βάλλη, η FTD. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Έχω μια ερώτηση, Πρόεδρε Ντράγκη, σε σχέση με μια ερώτηση που σας έχουμε αποστείλει γραπτός με τους αδέλφους. Μας δώσατε και μια απάντηση πριν από μερικές εβδομάδες, προσέλκυσε και τον ενδιαφέρον των μέσων Μεσικής ενημέρωσης. Με την απάντηση σας λοιπόν είπατε ότι αν τυχόν ένα νόμισμα έβγαινε από το ενίο νόμισμα, αν ένα κράτος έβγαινε από, την ενία, ε, από το ενιαίο νόμισμα θα έπρεπε να περάσει σε ένα διαφορετικό σύστημα ρύθμισης των ε, χρεών και των μισμάτων. Άρα ο τύπος ερμήνευσε αυτές τις δηλώσεις σας ότι εσείς δίνετε τη δυνατότητα της αναστρεψιμότητας του ευρώ, πράγμα το οποίο με αυτό δεν είχε ποτέ αναγνωριστεί ρητά από σας. Και άρα δίνατε την εντύπωση ότι θα έπρεπε σε μια περίπτωση εξόδου του ευρώ ότι ε, θα έπρεπε η Ιταλία να επιστρέψει 350 δισεκατομμύρια ευρώ ε, στην κεντρική τράπεζα, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ε, λόγω παθητικών πιστώσεων. Πώς όμως αυτά τα ποσά μπορούν να εντοπιστούν ως χρέος, να χαρακτηριστούν ως χρέος έναντι της ΕΚΤ και με ποια νομική βάση ή δεσμευτικά νομοθετήματα θα μπορούσε να ε, ζητήσει, να απαιτήσει την αποπληρωμή των ποσών αυτών η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πρόκειται για πιστώσει, δεν πρόκειται για στην πραγματικότητα για χρέο. Άρα θα ήθελα να ξέρω πού το στηρίζετε όλο αυτό που είπατε. Και έχω και άλλη μία ε, ερώτηση μετά την συνάντηση των σύπεδο αρχηγών κυβερνήσεων στη Μάλτα και με βάση και την έκθεση των πέντε ε, προέδρων που ανοίγει λίγο πολύ ένα σενάριο μεταρρύθμιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη δυνατότητα από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, χώρες όπως Φερρυπίνη, η Ελλάδα, η Ιταλία ή άλλες, ε, άλλες χώρες να μπορούσαν να βγουν για μια περίοδο από την Ευρωζώνη. Σε αυτή την περίπτωση και αν τυχόν πιέζει προς την διακατεύθυνση και η πολιτική, πώς θα δικαιολογούσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την έξοδο πρώτα και μετά την επανείσοδο στο ευρώ μιας χώρας. Απάντηση. Για την πρώτη σας ερώτηση θα απαντήσω λέγοντας ότι το ευρώ είναι μη αναστρέψιμο, ανέκλητο. Αυτή είναι η συνθήκη. This is the treaty. Και η απάντησή μου στην επιστολή σας ήταν απάντηση σε ένα τεχνικής φύσεως ερώτημα στηριζόμενο σε μια υπόθεση που δεν προβλέπουν οι συνθήκες αγγλικά. Και ως εκ τούτου η απάντησή μου στην ερώτησή σας, στην επιστολή σας, είχε να κάνει με ένα τεχνικό ζήτημα στηριζόμενο σε κυρώσεις που δεν προβλέπονται από τη συνθήκη. Σε υποθέσεις που δεν, δεν προέρχονται από τη συνθήκη. Για τη δεύτερη ερώτηση. Είναι πολύ πρόωρο να γίνει τέτοια κουβέντα. Δεν νομίζω ότι είναι σαφές αυτό που υπόθηκε στη Σύνοδο Κορυφής της Μάλτας. Έγινε λόγος για Ευρωπαϊκή Ένωση δύο ταχυτήτων, χωρίς όμως να είναι σαφές το ποιος, με ποιον τρόπο, πότε κτλ. Και δεν είχε αναπτυχθεί αυτή η ιδέα. Και άρα Πρόκειται μόνο για ένα σκαρίφημα θεώρηση ε, πάνω στο οποίο εγώ δεν μπορώ να κάνω κανένα σχόλιο σε αυτό το στάδιο. Μία ερώτηση μόνο ακόμη για το τεχνικό αυτό ερώτημα. Για το ποιε πιστώσεις θα μπορούσαν να συνιστούν χρέο και σε τι Αν θέλετε μπορούμε να απαντήσετε και γραπτός αν ε, σας εξυπηρετεί. Αλλά θα ήθελα μια απάντηση για την ερώτηση αυτή. Γιατί είναι ένα ζήτημα και ακαδημαϊκό θα έλεγα που έχει ανοίξει λίγο πολύ σε όλη την Ευρώπη. Απάντηση. Όπως έλεγα και πριν. Δεν θέλω να δώσω απάντηση σε μια ερώτηση στηριζόμενη σε υπόθεση που δεν προβλέπει η συνθήκη. Αυτό μπορώ να πράξω να σας αποστείλω γραπτή απάντηση μέσα στην οποία μπορώ να περιγράψω τις διαφορές μεταξύ του δικού μας συστήματος του Αρκεδίου και του συστήματος της Federal Reserve της ε, Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ. Επαναλαμβάνω στα αγγλικά, δεν μπορώ να δώσω απάντηση πάνω σε υποθέσεις στηριζόμενες ε, σε, βάση που δεν προβλέπεται στη συνθήκη, αλλά μπορώ να σας δώσω μία απάντηση γραπτή που θα κάνει τη διαφοροποίηση μεταξύ του δικού μας σύστημα, ε, συστήματος και της, ε, του συστήματος Federal Reserve. Καμπριέλ Μάτα, ευχαριστώ και ευχαριστώ κύριε Ντράγκη. Χαίρομαι. Ιδιαίτερω είμαι νέο μέλο στην Επιτροπή ΕΚΟΝ και νιώθω ιδιαίτερη χαρά. Όπω είπατε, το 2017 άνοιξε με θετικά στοιχεία, με τον πληθωρισμό να πλησιάζει στο 2%, το στόχο δηλαδή τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και επίση η ανάπτυξη φαίνεται ότι ε, παγιώνεται το δεύτερο εξάμεινο του 2016. Ε, η ΕΚΤ, ε, μάλιστα και η ΦΕΔ και η Κινέζικη Κεντρική Τράπεζα μείωσαν τις, τα μεσοπρόθεσμα επιτοκιά τους. Πιστεύετε ότι όλα αυτά θα μπορούσαν να... Η, πολιτική σας θα μπορούσε να είναι βάση και οδηγός και για άλλες κεντρικές τράπεζες και ποιο θα είναι ο αντίκτυπό ε, ε, του στι αγορέ του χρέου. Επίση, το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών την περασμένη εβδομάδα έδωσε στον πρόεδρο τη Federal Reserve μία επιστολή, στην οποία είναι σαφέ ε, το μήνυμα του Προέδρου ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στα αμερικανικά συμφέροντα σε όλε τι διεθνεί διαπραγματεύσει. Και σίγουρα αυτή δεν είναι καθόλου εύκολη ερώτηση. Η ερώτηση μάλλον είναι εύκολη, η απάντηση θα είναι δύσκολη σε τι φάση βρίσκονται οι σχέσεις σας με τη Federal Reserve, την Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα και τι προσδοκάται από την νέα Αμερικανική κυβέρνηση. Επίσης, σε ό,τι αφορά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Τραπεζών, της ΕΑΤ για την πιθανή ε, ίδρυση μιας κακιάς τράπεζας ε, που ε, θα συσσωρεύει τα κόκκινα δάνεια, δάνεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι περίπου ένα τρισεκατομμύριο ευρώ αυτά τα κόκκινα, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Ε, την περασμένη εβδομάδα σε μια διάσκεψη αναφέρθηκε η πρόταση ότι μια τέτοια κακή τράπεζα θα μπορούσε να βελτιώσει τους ισολογισμούς των τραπεζών απορροφώντας τα κόκκινα δάνεια. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση για την ίδρυση μιας τέτοιας κακιάς τράπεζας. Επίσης θα πρέπει να είναι μια ενιαία τράπεζα σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή κάθε κράτος θα πρέπει να έχει τη δική του κακιά τράπεζα που θα σωρεύει αυτά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Σε ό,τι αφορά την πρώτη σας ερώτηση για την επιστολή που εστάλει από το, κάποια μέλη του Αμερικανικού Κογκρέσου στην πρόεδρο της ε, Federal Reserve. Δεν πρόκειται εγώ ε, να σχολιάσω τι κάνει ένας ε, βουλευτής ή μέλος άλλης δικαιοδοσίας. Πάντως, αν με ρωτούσε, μου έστειλε κανείς παρόμοια επιστολή, θα μπορούσα να σας πω τι θα έλεγα εγώ. Νομίζω ότι όλοι μπορούμε να υποφεληθούμε από την ύπαρξη κεντρικών τραπεζών, εποπτών και ρυθμιστικών αρχών, γιατί οι μεγάλες οικονομίες μπορούν να μοιραστούν τις εμπειρίες τους από τις εποπτικές προδιαγραφές και μετά από δημόσιες διαβουλεύσεις. Τα τελευταία 30-40 χρόνια τέτοιου είδου διαβουλεύσεις, τέτοιες ανταλλαγές απόψεων ήταν πολύ θετικές και είχαν ε, ευνοϊκότατα αποτελέσματα. Και αυτές οι, διαβουλευσει είναι η αιτία της πρόσφατης ενίσχυσης του χρηματοπιστωτικού μας συστήματος με ένα πολύ πιο στεναρό ρυθμιστικό και αποπτικό πλαίσιο. Και μάλιστα δεδομένη της περιπλοκότητας ε, των παγκόσμιων αλληλεπιδράσεων μεταξύ των διαφόρων θεσμικών οργάνων. Σίγουρα είναι αναγκαίες τέτοιες ε, ανταλλαγές και συζητήσεις. Επί τη ευκαιρία, οι ρυθμιστικές και οι αποπτικές αρχές δεν δρουν απομονωμένα, ιδιαίτερα στο σημερινό κόσμο που όλα είναι αλληλένδετα. Τώρα, οι οι ρυθμιστικές αρχές, οι αποπτικές αρχές, οι κεντρικές τράπεζες έχουν τον τελικό λόγο για τη για το αριθμιστικό πλαίσιο ή την ε, χρηματοοικονομική χρηματοπιστωτική νομοθεσία. Όχι βέβαια, ούτε εδώ, ούτε στι Ηνωμένε Πολιτείε, ούτε και πουθενά άλλου. Πάντα οι νομοθέτε έχουν το λόγο, όχι τον τελικό αλλά και τον αρχικό. Έχουν την φυσιολογική διακριτική ευχέρεια να εφαρμόσουν τις απόψεις που συζητήθηκαν μετά από διαβουλεύσεις με τις ρυθμιστικές αρχές, εποπτικές αρχές και τις κεντρικές τράπεζες. Αλλά οι νομοθέτες έχουν το λόγο τελικά. Οπότε αυτό θα παντούσαν λάβανα παρόμοια επιστολή. Τώρα, σε ό,τι αφορά το δεύτερο σας σχόλιο, την ίδρυση μιας κακής τράπεζας ή μιας εταιρείας διαχείρισης στοιχείων του ενεργητικού για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, NPL, τέτοιου είδους εταιρείε διαχείρισης εκφύσεως είναι περίπλοκης δομής και το διαπιστώσαμε και το βιώσαμε στο πρόσφατο παρελθόν και μάλιστα επανειλημμένος. Ακόμη πιο περίπλοκο θα ήταν μια εταιρεία διαχείρισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης θα πρέπει να διαρωτηθούμε, μια εταιρεία διαχείρισης αυτές οι κακές τράπεζες, θα είναι πανάκια για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, για τα κόκκινα δάνεια. Η απάντηση είναι όχι βέβαια, μάλλον όχι. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τα δύναμα στοιχεία του ενεργητικού ή τα κακής ποιότητα στοιχεία του ενεργητικού θα έπρεπε να αντιμετωπιστούν με ρηξικέλευθες αλλαγές στο νομικό ε, δικαστικό και ρυθμιστικό κανονιστικό πλαίσιο και πρώτα απ' όλα σε εθνικό επίπεδο. Για παράδειγμα, διαδικασίες για την ανάκτηση του χρέους, εξοδικαστικές διευθετήσεις ή διακανονισμοί, η δημιουργία μιας αγοράς για τα κόκκινα δάνεια, για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Όλα αυτά είναι απαραίτητα στοιχεία της αντιμετώπισης του προβλήματος. Η ίδρυση μιας εταιρείας διαχείρισης είναι ίσως ένα μόνο από τα πολλά μέτρα που θα χρειαστεί να ληφθούν για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Σας ευχαριστώ. Thank you. Ε, ευχαριστώ πολύ, η Νίνα Τζιλ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Ντράγκη, πολύ σωστά είπατε ότι Βλέπουμε επιτέλους ε, ανάκαμψη στην Ευρώπη. Θετική είναι η προοπτική για την οικονομία και σίγουρα αξίζετε και εσείς ε, τα εύσημα για, από πλευράς ΕΚΤ. Όμως, σε ό,τι αφορά αυτή την ανάκαμψη, θα σα πω πρώτα ότι στι 10 Ιανουαρίου γράψατε στο συντονιστή μου μια επιστολή και εκφράσετε την ανησυχία σας για το Brexit, ότι μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια εποπτείας ε, τη ΕΚΤΑ στα Βρετανικά τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και είπα ότι είναι σημαντικό να βρεθούν λύσεις που στην ε, ε, καλύτερη περίπτωση θα βελτιώσουν, στη χειρότερη θα διατηρήσουν ε, το στάτους quo σε ό,τι αφορά την εποπτεία. Σε ό,τι αφορά όμως ε, ε, την καθάριση κάποιων προϊόντων ε, υπηρεσιών στην Ευρωζώνη, μπορεί αυτό να επηρεάσει. Γιατί κάποια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δεν θα μπορούν να συνεισφέρουν στην καινοτομία, την ανάπτυξη, τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας. Ότι Μάσαρτ και άλλοι υπερογνώμονες ανησυχούν μήπως με μια περιοριστική τέτοια πολιτική συμψηφισμού, clearing, θα επηρεαστούν αρνητικά. Όσοι έχουν ένα συνταξιδοτικό πρόγραμμα, κάποιο επενδυτικό συμμετέχουν, θα είναι δηλαδή μια κατάσταση από όπου θα βγουν όλοι χαμένοι. Μια δραστική πολιτική μετεγκατάσταση. Έχει και ένα κίνδυνο. Μπορεί να υπάρξουν αντίπεινα από άλλες χώρες και να επηρεάσει αυτό τα χρηματοπιστωτικά δρήματα που έχουν την έδρα τους ε, στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο όταν απαντήσατε, είπατε ότι θα πρέπει να έχει ένα ρόλο η ΕΚΤ στους κεντρικούς αντισυμβαλόμενους. Θα μπορούσε να υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ ΕΚΤΑ και Τράπεζα της Αγγλίας. Αυτό νομίζω ότι θα επέτρεπε να συνεχίσει να πτήσεται η ευρωπαϊκή οικονομία. Δεύτερο σημείο για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Βέβαια, απαντήσατε στα περισσότερα ερωτήματα. Πέντε δευτερόλεπτα έχετε ακόμα. Μάλιστα. Εγώ ανησυχώ. Αυτό το οποίο προτείνετε, μήπω ε, πάρει πολύ χρόνο, δεν υπάρχει ένα πιο γρήγορο τρόπο να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Thank you. right now, the... E Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή η ΕΚΤΑ συμμετέχει στην εποπτεία των κεντρικών αντισυμβαλόμενων στη Βρετανία μέσω των εποπτικών αρχών που έχουν δεσπιστεί από το ΕΜΡ. Και υπάρχει και ένα μνημόνιο συνεννόηση με την Τράπεζα της Αγγλίας, ειδικά για το θέμα αυτό. Η συνεργασία μας με την Τράπεζα της Αγγλίας και ασφάλεια δικαίου που προσφέρει και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Υπάρχει ένα πλαίσιο λοιπόν. Αυτό το πλαίσιο μας επιτρέπει να παρακολουθούμε τους κινδύνους στο νομισμά μας είναι πολύ νωρί, θα σα έλεγα, να τοποθετηθούμε ξεκάθαρα πάνω στο ρυθμιστικό πλαίσιο που θα πρέπει να εγκαθιδρυθεί όταν θα εγκαταλείψει την Ένωση το Ηνωμένο Βασίλειο. Βασική μα ανησυχία θα είναι η χρηματοπιστωτική σταθερότητα, η προστασία των επενδυτών και βέβαια το ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού για τους καταναλωτές, τους πολίτες και τις εταιρείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θα είναι ο στόχος μας. Ιδίω αυτό που είναι σημαντικό είναι να μην επαναχωρήσουμε σε ό,τι αφορά την ενιαία αγορά. Αν κάποιο θέλει να είναι στην ενιαία αγορά, σημαίνει ότι είναι, υπάγεται, υπόκειται στο, ε, στη δικαιοδοσία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα, αλλά επαναλαμβάνω είναι πολύ νωρί για να πούμε κάτι πιο συγκεκριμένο. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο σα ερώτημα, για το κατά πόσο θα υπήρχε ένα πιο γρήγορο τρόπο για την αντιμετώπιση του προβλήματο των μη εξυπηρετούμενων δανείων, δυστυχώ δεν υπάρχει είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους ε, τόσο καιρό επιμένει αυτό το πρόβλημα. Σίγουρα αποτελεί μείζωνα πρόκληση για κάποιες ευρωπαϊκές τράπεζες και για ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες. Είναι και ένας από τους βασικούς παράγοντες που, που κρατούν την κερδοφορία των ορισμένων τραπεζών σε χαμηλά επίπεδα. Φυσικά όταν έχουμε χαμηλούς συντελεστέ, χαμηλή ανάπτυξη, όλα αυτά ε, επηρεάζουν. Και στον τομέα ε, υπάρχει ένα είδος συνοστισμού, αν μπορώ να το χαρακτηρίσω έτσι, που και αυτό επηρεάζει το κληροδότημα, αυτή η κληρονομιά αυτών των πολλών μη εξυπηρετούμενων δανείων ε, έχει μειώσει την κερδοφορία των τραπεζών και έχει μειώσει την ε, ε, δυνατότητα δράσης τους. Αυτό που χρειάζεται λοιπόν είναι μια στρατηγική όπου εθνικές μεταρρυθμίσεις, στους το που δικαστικό τομέα, νομικό τομέα, ρυθμιστικό τομέα, είναι κάτι απαραίτητο και ιδίω ό,τι αφορά τα τοξικά δάνεια, που είναι ακριβώ κληροδοτημένα το να ε, εισαγάγουμε νέα νομοθεσία. Δεν βοηθάει ιδιαίτερα, γιατί πώ θα αντιμετωπίσουμε τα προϋπάρχοντα αυτά τοξικά δάνεια, με εξυπηρετούμενα δάνεια. Πρέπει να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Βλέποντας δε ότι η βελτίωση στις οικονομικές συνθήκες ε, συνολικά ήταν ευνοϊκή για την κατάσταση. Βλέπουμε ότι είναι λιγότερα, είναι μειώνονται τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια λόγω της βελτίωσης των οικονομικών συνθήκων. Και σε ό,τι αφορά τον νέο μηχανισμό και την ΕΚΤ, ξέρετε ότι θα δημοσιεύσουμε για δημόσια διαβούλευση σχέδιο κατευθυντηρίων γραμμών για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια φέτος ε, στις αρχές του έτους θα δημοσιοποιηθεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ η Χούμπνερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Ντράγκη, έχω ένα ερώτημα σε σχέση με τη ρευστότητα των αγορών και στο πλαίσιο με ενδεχόμενη ε, εξομάλυσης πολιτικό, γιατί πολλές φορές ε, οι κλάδοι, οι βιομηχανίε παραπονούνται, εκφράζουν την ανησυχία τους λόγω νέων στοιχείων αυτού του ε, νέου πλαισίου, MIFID, EU κτλ. Ε, ότι θα δημιουργήσει κάποια προβλήματα, ιδίως για το, σε σχέση με το ότι οι τράπεζες αποσύρονται από δραστηριότητες που γεννούν χρήμα ουσιαστικά και δεν έχουν πιστεί. Το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης έχει δώσει πολύ ρευστότητα που ίσως να συγκαλύπτει κάποια προβλήματα, τα οποία όμως θα επαναναδυθούν όταν εξομαλυνθούν οι πολιτικές. Ερωτώ λοιπόν, παρακολουθείτε τον αντίκτυπο του ρυθμιστικού πλαισίου σε ό,τι αφορά τη ρευστότητα. Είναι κάτι το οποίο λαμβάνεται υπόψη. Και τι είδους τοπίο αν μπορώ να το πω έτσι, περιμένετε ε, για τη ρευστότητα όταν ε, πλέον έχετε χάραξη στρατηγική εξόδου. Το Δεκέμβριο ε, από το ESRB ακούσαμε ότι σκέφτονται για ένα νέο φορέα και συγκεκριμένα για τα ομόλογα, τα κρατικά και εκεί προβλέπεται ένας επιμερισμός ε, των κινδύνων. Υπάρχει και ένα θέμα όμως ότι αυτή η τίτλη, τα αξιόγραφα είναι πολύ πιο πολύπλοκα προϊόντα και πολύ λιγότερο ρευστά από τα κρατικά ομόλογα και θα πρέπει να δούμε το κατά πόσο θα είναι για τους επενδυτές, αν θα βρουν αγορές ε, υπάρχει ένα ενδεχόμενο ανταγωνισμό μεταξύ των νέων χρεογράφων και αυτών που κάνει μέχρι στιγμή η ΕΚΤΑ κρατικά ομόλογα, δηλαδή αγορά κρατικών ομολόγων. Θα μπορούσατε να τα σχολιάσετε αυτά. Ευχαριστώ. Θα απαντήσω πρώτα, στο δεύτερο ερώτημα. Είμαστε σε πολύ πρόημο στάδιο ακόμη Την προσπάθεια αυτή δεν ε, την καθοδηγεί η ΕΚΤΑ. Ουσιαστικά περί τίνος πρόκειται. Υπάρχει μια task force στο ESRB, δηλαδή το Συμβουλίο Συστημικού Κινδύνου. Και εκεί εκπροσωπούνται όλοι οι διοικητές των κεντρικών τραπεζών που προσπαθούν να βρουν αυτά τα ασφαλή ομόλογα, τα ασφαλή ευρωπαϊκά ομόλογα. Θα δούμε τι θα προκύψει από το έργο αυτής της ομάδας εργασίας. Μέχρι στιγμής τι γνωρίζουμε, ότι ουσιαστικά βασίζεται 100% το από αυτό στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έχουν ευθύνε οι εθνικέ κυβερνήσει σε ό,τι αφορά την έκδοση, για παράδειγμα, τη βιωσιμότητα του χρέου ή την ε, εξυπηρέτηση του χρέους. Ουσιαστικά λοιπόν είναι κάτι το οποίο ακόμη μια πολύ πρόημο να σχολιάσει κανείς. Ειλικρινώς δεν μας έχει καν απασχολήσει το ερώτημα ακριβώς όπως το θέτετε εσείς, τι θα γίνει με τα κρατικά ομόλογα κτλ. Διότι ακόμη δεν έχει φτάσει σε αυτή τη φάση το όλο ζήτημα. Σε ό,τι ρευστότητα, το άλλο σας ερώτημα. Εν γέννη και ανεξαρτήτως αλλαγών των κανονισμών, η έξοδος από μια παρατεταμένη περίοδο πολύ επεκτατική νομισματική πολιτική και αρνητικών, τέλο πάντων πολύ χαμηλών επιτοκίων, είναι κάτι που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή για πολλού λόγου. Ένα από του οποίου είναι το γεγονό πω ε, οι συμμετέχοντε ε, στην αγορά μόλι έχουν προσαρμοστεί ε, για αυτή την, σε αυτή την κατάσταση, τη ρευστότητα δηλαδή. Μέχρι στιγμής δεν βλέπουμε πρόβλημα έλλειψη ρευστότητας Ίσως σε μικρά τμήματα της αγοράς να παρατηρείτε κάτι τέτοιο. Αλλά γενικά δεν παρατηρούμε έλλειψη ρευστότητα. Φυσικά βέβαια και θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και να παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς ε, το ζήτημα αυτό, διότι έχουμε την εμπειρία από την κρίση και από άλλες περιπτώσεις ότι η ρευστότητα υπάρχει όσο υπάρχει. Έρχεται και φεύγει και πολύ εύκολα εξαφανίζεται. Εξού ορισμένα ρυθμιστικά μέτρα θα εφαρμοστούν ακριβώς για να αποφευθούν ευνίδι, κλειδονισμοί και αλλαγές με την ρευστότητα ή για να εξασφαλιστεί ανθεκτικότητα σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο Πέντρο Σίλβα Περέιρα. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, μας ε, εκθέσατε πολύ πιστικά επιχειρήματα στην ομιλία σας ε, για να τεκμηριώσετε την ανάγκη της συνέχισης αυτής της διευκολυντικής πολιτικής ε, και επεκτατικής νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με μη συμβατικά μέτρα. Αυτή που ζητούν από την Ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα μία ρηξικέλευτη και ευνίδια αλλαγή, μια πιο περιοριστική δηλαδή πολιτική, φαίνεται ότι κάνει μια πολύ κακή εκτίμηση, εσφαλμένη εκτίμηση της ευρωπαϊκής οικονομίας και σκέφτονται περισσότερο τα δικά του συμφέροντα παρά τα συμφέροντα του συνόλου της Ευρωζώνης. Και όπως είπατε και εσείς σε άλλη περίπτωση, θα πρέπει να δείξουν εμπιστοσύνη και υπομονή πρώτα απ' όλα, να έχουν υπομονή. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δράγκη, τονίσατε στην ομιλία σας την ανάγκη της σύγκλησης. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω αν αναγνωρίζετε ή όχι ότι στις πρόσφατες αλλαγές της νομισματικής πολιτικής και ιδιαίτερα στα κριτήρια του προγράμματος αγοράς περιουσιακών στοιχείων, αν ε, υιοθετήθηκε μία λύση που είχε ασύμετρα αποτελέσματα στην Ευρωζώνη. Δηλαδή ήταν μια λύση που ευνόησε μερικούς εις βάρος κάποιων άλλων όμως. Για παράδειγμα, έκανα τις επενδύσεις ε, στο γερμανικό χρέος ε, πολύ πιο ελκυστικές και άρα πολύ λιγότερο ε, ελκυστικές έγιναν οι επενδύσεις προς το χρέος των περιφερειακών χωρών της Ευρωπαϊκής της Ευρωζώνης. Και αν ισχύει κάτι τέτοιο, σα απασχολεί αυτό το πρόβλημα, σας ανησυχεί καθόλου. Δηλαδή, δεν θα έπρεπε στην νομισματική σας πολιτική να ε, σκεφτείτε και κάποιους μηχανισμούς στήριξης, της σύγκλησης, ώστε να αποφύγουμε καταστάσεις που επιδεινώνουν τη σύγκληση ή επιτείνουν την απόκληση στην Ευρωζώνη. Και τέλος, θα ήθελα να ρωτήσω, αν στις χώρες που είχαμε ε, επίπεδο αγοράς περιουσιακών στοιχείων κάτω από το όριο που που προβλε... παρά όλο που λαμβάνουν την υπόψη και άλλες συνθήκες. Αυτές οι χώρες μπορούν να ελπίζουν σε μία επαναφορά σχετικά γρήγορα του κανονικού επίπεδου αγοράς, ώστε να μην ε, επιδεινωθεί η κατάσταση του χρέους τους και του κρατικού τους ομολόγου στις αγορές. Ευχαριστώ. θα πρέπει να έχουμε συνεχώς κατά νου ότι στόχος μας και η εντολή μας είναι να ε, καταλήξουμε σε μία σταθερότητα των τιμών και σε ένα ποσοστό πληθωρισμού που θα είναι ε, λίγο κάτω από το 2% μέσω πρόθεσμα. Και ε, ο, πολιτικός, ο προσανατολισμός της νομισματικής μας πολιτικής χαρακτηρίζεται από αυτό και σε ε, στόχος μας είναι ένα επίπεδο πληθωρισμού που θα ε, πληρεί τις τέσσερις προϋποθέσεις που σας ανέφερα προηγουμένως, τα τέσσερα χαρακτηριστικά. Και γι' αυτό ε, εγκρίναμε το πρόγραμμα των αγορών και μάλιστα κάναμε κάποιες αλλαγές το Δεκέμβριο ώστε να αγοράσουμε κάτω από τη δυνατότητα καταθέσεων και μάλιστα το Διοικητικό Συμβουλίο στις τελευταίες συνεδρίες εξέφρασε την ικανοποίησή του για τα αποτελέσματα της απόφασης του Δεκεμβρίου. Και μάλιστα, όπως είπα και προηγουμένως, διαπιστώσαμε ότι η νομισματική μας πολιτική συνέβαλε στη βελτίωση και στην παγίωση της ανάκαμψης που παρατηρούμε σήμερα και σε βελτιωμένες συνθήκες και στην αγορά εργασίας και μάλιστα έθεσε τις προϋποθέσεις για την βελτίωση και του βασικού πληθωρισμού, πέραν της ε, αύξησης του γενικού πληθωρισμού που οφείλεται και σε αλλαγές της, ε, ε, στη τιμή της ενέργειας και τα αποτελέσματα που είχαν. Τώρα, κατά τη διεξαγωγή αυτού του προγράμματος αγορών, είναι σαφές ότι δεσμευόμαστε όχι μόνο από την κλίδα κεφαλαίου, capital key, αλλά και από αυτό που είπα προηγουμένως, το όριο έκδοσης και το όριο εκδότη. Και ο λόγος των ορίων αυτών είναι ότι θέλουμε να φροντίσουμε ότι δεν θέλουμε να εφαρμόσουμε κάποιες παρατηρήσεις εποπτεία των των χρηματαγορών, κάτι που απογορεύεται από τη συνθήκη και θέλουμε να αφήσουμε τις ε, αγορές να λειτουργήσουν. Αν θέλουμε να αγοράσουμε ένα μεγαλύτερο μερίδιο του δημόσιου χρέους μιας ε, αλφα χώρας, κατά πάσα πιθανότητα θα, αντιτα... θα καταπατήσουμε αυτά τα δύο κριτήρια. Δηλαδή, θα δοθεί εντύπωση ότι πραγματοποιούμε αυτό το monitor financing και επίσης ε, θα θεωρηθεί ότι οι, ενέργειες μας, οι διαστρεβλώνουν τη λειτουργία της αγοράς υπέρ μιας χώρας. Γι' αυτό και ορίσαμε όρια και έκδοσης και εκδότη. Οπότε δεν ε, νομίζω ότι η, το πρόγραμμα αγοράς οδηγεί σε ανισότητα. Ευχαριστώ, Βέρνερ Λάγκεν. Πρόεδρε. στις 28 Νοεμβρίου είπατε ότι είναι σημάδια κρίσης στα χαμηλά επιτόκια. Και ταυτόχρονα δώσατε μια θετική αξιολόγηση για τα συνολικά επιτόκια στην Ευρωζώνη. Τώρα βλέπουμε προ το παρόν μια αντίστροφη τάση. Το spread έχει γίνει μεγαλύτερο, ιδιαίτερα μεταξύ Γερμανίας, Ιταλία, αλλά και έναντι άλλων κρατών. Άρα είναι όλο και μεγαλύτερη η απόσταση στα spread. Ε, ο πληθωρισμός σε αρκετές χώρες ε, είναι πολύ κάτω από το 2% και εκεί που είναι οι περισσότεροι επενδυτές παραδοσιακά παραμένουν πολύ χαμηλά τα επιτόκια. Πολύ χαμηλά. Άρα λοιπόν κάποια στιγμή θα πρέπει, άπαξ και αρχίσουν να ανεβαίνουν και τα επιτόκια στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον χώρο του δολαρίου, να προχωρήσετε κι εσείς αντίστοιχες ορθωτικές κινήσεις. Προς το παρόν όμως βλέπουμε κάτι το αντίστροφο να συμβαίνει με την επέκταση του προγράμματός σας και βλέπουμε η κατάσταση να έχει φτάσει μέχρι το σημείο αυτό από τον Νοέμβριο που είμαι αναγκασμένος να ρωτήσω Πώς βλέπετε το μέλλον όταν έχουμε τόσο μαζικές αλλαγές στους τελευταίους μήνες. Δεύτερη ερώτηση. Έχει πει αλλά έχει ταυτόχρονα και υπογράψει διάταγμα ο πρόεδρος Τραμπ σε σχέση με την ανατροπή ε, κανονιστικών ρυθμίσεων, αλλά έχει κάνει και δηλώσεις που θα οδηγήσουν στην ανατροπή της ίδιας της Σύμβασης της Βασιλείας. Και επίσης, μετά από τα 25 χρόνια της συνθήκης του Μαστρίχτ και την υπογραφή από εσά της έκθεσης των πέντε προέδρων, τι είδου ε, μέτρα θα κρίνατε εσείς και ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ως εκ των φόρους για να ε, προχωρήσει αυτή η... ο πρόεδρος. Ο κύριος Στράικη, με συγχωρείτε, ε, ποια ήταν η τελευταία σας ερώτηση σε σχέση 25 χρόνια Μάστριχτ, λέει ο κύριος Λάγκε, και θεσμικές μεταρρυθμίσεις τι έχετε να προτείνετε. Και με βάση βέβαια και την έκθεση των πέντε πρόεδρων. Ο κύριος Δράκη. Για την πρώτη ερώτηση. Έχουμε υποστεί επικρίσει από διάφορε πλευρέ στην Ευρωζώνη, γιατί είναι νομισματική η πολιτική μας βέβαια, η οποία λένε ε, μπορεί να ανατρέψει την ε, πειθαρχία των αγορών. Βλέπουμε όμως ότι δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αντιδρούν οι αγορές όντως. Αλλά αντιδρούν σε διαφορετικές συνθήκες. Διάφορες συνθήκες. Και εδώ εγώ θα συνιστούσα να προωθούνται και οι δημοσιονομικές πολιτικές σε όλες τις χώρες κατά τρόπο ώστε να ευνοούν την ανάκαμψη. Ανάκαμψη βιώσιμη ταυτόχρονα. Άρα, χώρες οι οποίες δεν έχουν δημοσιονομικό περιθώριο δεν θα πρέπει να προσπαθούν να το εξαντλούν πιεστικά δηλαδή να προχωρούν στην εξέβρεση δημοσιονομικού περιθωρίου όταν αυτό δεν υφίσταται. Αντίθετα θα πρέπει να προχωρούν σε μια διαφορετική διατύπωση, σύσταση του προπολογισμού. Και το έχουμε πει πολλέ φορέ ότι αυτοί οι προπολογισμοί τη γενική κυβέρνηση θα πρέπει να διαμορφωθούν κατά τρόπον ευνοϊκό στην ανάπτυξη. Και άλλωστε το έχουμε πει και αυτό, είναι απαραίτητο να αλλάξει η σύνθεση του προπολογισμού, αλλά ταυτόχρονα και να γίνουν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Η ερώτηση σας, η δεύτερη, ε, ε, αναφερόταν στο ε, πότε θα αλλάξουμε στάση exit. Την ίδια απάντηση που έδωσα και νωρίτερα θα σας δώσω. Ο στόχος μας είναι το ποσοστό του πληθωρισμού, το οποίο είναι κοντά, αλλά κάτω από το 2% μέσω πρόθεσμα. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που σας κάνει να γελάτε. Έστω. Πρέπει λοιπόν ε, να είμαστε και πεπισμένοι πως είναι ε, σταθερά συγκλίνοντας οι στόχοι αυτοί. Παρακολουθούμε λοιπόν τις τάσεις εξελίξεων στον ονομαστικό πληθωρισμό. Και επίσης, όπως είπα, πρέπει να ισχύει για όλη την Ευρωζώνη και να είναι αυτόνομα αηφόρος βιώσιμος. Αυτές είναι οι προοπτικές για την αλλαγή της στάσης μας στην νομισματική πολιτική. Για τη δεύτερη ερώτηση και την χρηματοοικονομική απορρίθμιση. Όπως είπα και νωρίτερα, πρέπει να μπορέσουμε να εξετάσουμε με ακρίβεια αυτό που προτίθεται να πράξει η κυβέρνηση των ΗΠΑ σε σχέση με την ε, Σύμβαση Βασιλεία 3, η οποία μέχρι ενός μηνός, μέχρι όσο μηνός ίσχυε και λειτουργούσε με την προηγούμενη, την απερχόμενη κυβέρνηση, ναι, μάλλον κυβέρνηση των ΗΠΑ. Πρέπει να δούμε λοιπόν τι ακριβώς θα προκύψει στο μέλλον. Αλλά πάντως, και το επαναλαμβάνω, ο συνδυασμός της ποσοτικής χαλάρωσης και της χρηματοοικονομικής απορρίθμισης ήταν ακριβώς η βάση πάνω στην οποία στηρίχθηκε και ανεπτύχθη η χρηματοοικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση και, τι είναι δεδομένη η υφιστάμενη επεκτατική νομισματική πολιτική με στόχο την επίτευξη του στόχου μας, με πάσα ειλικρίνα σας λέγω ότι δεν βλέπω κανένα λόγο για χαλάρωση του υφισταμένου ρυθμιστικού πλαισίου, αυτού το οποίο έχει οδηγήσει σε μια πολύ πιο στεναρή σε ένα πολύ πιο στεναρό τραπεζικό περιβάλλον και γενικότερα χρηματοοικονομικό περιβάλλον από ό,τι είχε συμβεί στο παρελθόν με άλλες πολιτικές. Επίσης αναφέρεστε σε θεσμικές αλλαγέ. Υπάρχει όμω όχι ένα σκαρίφημα, υπάρχει ένα σαφέ σχέδιο οδικός χάρτης ή φιλοπορίας που προκύπτει από την έκθεση των πέντε προέδρων και νομίζω ότι είναι σαφές και πρέπει να είναι σαφές για τους πάντες πως έχουμε δύο άξονες πολιτικής δράσης που πρέπει να αναπτυχθούν. Ο πρώτος σε εθνικό επίπεδο και σημαίνει ότι πρέπει να συγκλίνουν περισσότερο οι οικονομίες μας. Μια προϋπόθεση άλλωστε, μια υπόθεση την οποία είχαν υπόψη εκείνοι οι οποίοι υποστήριξαν τη συνθήκη του Μανστρίχτ, ότι δηλαδή θα, γίνει πραγματική, θα υπάρξει πραγματική σύγκληση. Η πραγματική σύγκληση μπορεί να γίνει με μεταρρυθμίσεις διαρθρωτικές. Δεύτερον, δεύτερος άξονας, την ίδια χρονική στιγμή ή αμέσω μετά το σύμφωνο, την συνθήκη του Μαστρίχτη, είχαμε το σύμφωνο σταθερότητα και ανάπτυξη. Δηλαδή την τήρηση των κανόνων. Με την σύγκληση και την τήρηση των κανόνων μπορούμε να οικοδομήσουμε αυτή τη βάση εμπιστοσύνης η οποία θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε με βαθύτερη ευρωπαϊκή νομισματική ολοκλήρωση και τη δημιουργία των σχετικών θεσμών. Προχωρούμε λοιπόν κατά τρόπο παρόμοιο ουσιαστικά με τα όσα έχουν ε, γίνει για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Από διαφορετικές δηλαδή και χωριστές πολιτικές προχωρούμε σε μια ενοποιημένη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά βέβαια αυτό προϋποθέτει και εμπιστοσύνη. Ευχαριστώ, Φέρνατε Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ κύριε και καλώς ήλθατε. Τρεις ερωτήσεις θα ήθελα να σας πω πολύ γρήγορα. Στην πρώτη ερώτηση αναφέρθηκε ήδη η συνάδελφος Ντανούτα Χούπνερ για αυτή την πρόταση που φαίνεται ότι υποβάλλει η Κομισιόν μέσω του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κίνητου το οποίο προεδρεύετε εσείς, δηλαδή για την τιτλοποίηση δημόσιου χρέους. Εσείς είπατε ότι ακόμα είναι πρώιμο το στάδιο των εργασιών. Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Πότε περιμένουμε μια έτσι λίγο πολύ πιο επίσημη πρόταση. Πώς αξιολογείτε εσείς αυτές τις εργασίες. Θα ήθελα να μας δώσετε λίγο περισσότερες λεπτομέρειες για τη συζήτηση στο Συμβούλιο στην Κινδύνου. Το δεύτερο ερώτημα αφορά την έκθεση Μόντι για τους ίδιους πόρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως γνωρίζετε, εδώ και καιρό επιμένουμε για τη δυνατότητα να μπορεί για τις χώρες της Ευρωζώνης να υπάρχει αυτή η πρόβλεψη για, τη, για, τη, για τους ίδιους που περιλαμβάνεται και στην έκθεση Μόντι και σε ό,τι αφορά αυτό που είπε και ο Στάρφο Λάγκεν, τι απομένει να γίνει στη στο θεσμικό σχεδιασμό και σε σχέση πάντα με την 65 προέδρων, υπάρχουν καθυστερήσεις. Πώς τις αξιολογείτε. Υπάρχουν καθυστερήσεις στο Συμβούλιο για τη συζήτηση των εισφορών Λέβη. Ε, και σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου. Τι έχετε να μα πείτε. Για τα ομόλογα απάντησα και είπα ότι είναι πολύ νωρίς για να κάνουμε κάποιο σχόλιο. Δεν είναι κάτι ε, που εξετάζεται άμεσα από την ΕΚΤ. Όπως είπα υπάρχει σχετική ομάδα εργασίας Task Force. Ε, κεντρικός διοικητής ε, της Ιρλανδίας είναι ο αρμόδιος και προσωπούνται και όλες οι κεντρικές τράπεζες με τους διοικητές τους. Θα πρέπει να δούμε που θα καταλήξει η Task Force και μετά μπορούμε να την αξιολογήσουμε την πρόταση τη σχετική. Είναι σαφές ότι πρόκειται για 100% κόνσεπτ ιδιωτικού τομέα που όμως σημαίνει ότι οι κυβερνήσεις εξακολουθούν να έχουν ευθύνες ό,τι αφορά τη δημοσιονομική πολιτική, σε ό,τι αφορά την εξυπηρέτηση του χρέους, για παράδειγμα. για την επιστροφή ε, κερδών της ΕΚΤΑ στον κοινοτικό προπολισμό είναι κάτι το οποίο πονέστε με δεύτερη σα ερώτηση. Αυτό είναι μια πολιτική απόφαση για την οποία απαιτείται αλλαγή στη δομή, στο καταστατικό συγγνώμη του ΕΚΤΑ. Και γι' αυτό θεωρούμε ότι θα χρειαστεί και αλλαγή της συνθήκης. Και η έκθεση μόνη τη συμφωνεί Δεν μπορεί αυτό να γίνει στο πλαίσιο της αποστευμένης διαδικασίας. Το 33 ένα β για τη διανομή των αναπομεινών κερδών της ΕΚΤΕ. Είναι αυτό το άρθρο που θα πρέπει να ε, τροποποιηθεί. Ουσιαστικά προβλέπεται η κανονική διαδικασία να θεωρείται Το άρθρο 48 της συνθήκης προβλέπεται αυτό. Άρα, κατά την άποψή μας, αφισβητείτε το κατά πόσον με τροποποίηση του 33.1 ε, α για την ε, διανομή μέρους ή όλων των κερδών της έκτασης στον ευρωπαϊκό περιπολισμό με την απλοποιημένη διαδικασία είναι κάτι που από νομικής πλευράς ευσταθεί. I'm sorry? It was a question on, yeah, on Oh, I'm sorry. Κάνετε και ένα άλλο ερώτημα. Ουσιαστικά ο άλλο πυλώνα της ε, Τραπεζικής είναι το έτης και θα πρέπει να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Όπως είπα και πριν, είμαστε υπέρ μια παράλληλης προσέγγισης, δηλαδή μείωση κινδύνου, επιμερισμό κινδύνων. Ε, από πάντα είχαμε την προσέγγιση αυτή βέβαια και έχουν ληφθεί διάφορα μέτρα για τη μείωση των κινδύνων. TILAC, MRL, Net Stable Funding Ratio, Leverage Ratio. Πολλά μέτρα έχουν εφαρμοστεί. Ίσως και σε ό,τι αφορά την ενοποίηση του τραπεζικού τομέα και την ενίσχυσή του θα ήταν κάτι που θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε αλλά και τον επιμερισμό κινδύνων θα τον συνεχίσουμε. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστώ, Αλένα Μασού. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Μας υπενθυμίσατε, κύριε Πρόεδρε, ότι ένα από τα οξύμορα της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης είναι ότι η σύγκληση μεταξύ των οικονομιών της Ευρωζώνης μάλλον οπισθοδρόμησε από την κρίση κυρίως και μετά. Ένα άλλο ξύμορο είναι ότι από την εποχή της κρίσης διαπιστώνεται κατακαιρματισμός, διάλυση τη αγορά των κεφαλαίων, κάθε τράπεζα, κάθε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα δηλαδή, αναδιπλώνεται προς την εθνική της αγορά. Και αυτός ο κατακαιρματισμός διατηρείται ακόμη και σήμερα, πράγμα ιδιαίτερα ανησυχητικό. Κατά κάποιο τρόπο δηλαδή η ποσοτική χαλάρωση, η quantitative είναι κάτι θετικό βεβαίως, αλλά εμέσως είναι και ένας τρόπος να ενθαρρύνει αυτόν τον κατακαιρματισμό. Ε, πιστεύετε λοιπόν ότι για να επανέλθουμε στην ελεύθερη διακίνηση των κεφαλαίων και των, διασυνο... και, της... Ε, και των διασυνοριακών επενδύσεων από τράπεζες και άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς απαιτείται πρωταρχικά εμπιστοσύνη, αυτό είναι το κύριο πρόβλημα που επικαλεστήκατε και νωρίτερα ή υπάρχουν και προβλήματα σε σχέση με τον επιμερισμό των αρμοδιοτήτων μεταξύ του ρυθμιστικού ευρωπαϊκού δηλαδή επίπεδου και του εθνικού του. Ευχαριστώ. απάντηση. Η πρώτη παρατήρηση έχει να κάνει με τη σύγκληση των οικονομιών μας. Υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία που δείχνουν ότι η διασπορά της ανάπτυξης της προσθέμενης αξίας της χώρας της Ευρωζώνης έχει μειωθεί σημαντικά και βρίσκεται τώρα στο χαμηλότερο ιστορικά επίπεδο από την ε, έναρξη της κυκλοφορίας του ευρώ. Είμαι πεπισμένο λοιπόν ότι καθώ θα προχωρά και η ανάκαμψη πάλι θα συνεχίσει να μειώνεται αυτή η διασπορά. Έχω όμω και επανειλημμένα τονίσει ότι πρέπει αυτή η ανάπτυξη να είναι βιώσιμη και για να είναι αυτή βιώσιμη πρέπει να ε, περάσουν μέσα από τις ε, απαραίτητε μεταρρυθμίσει οι χώρε με βάση το εθνικό πρόγραμμα η καθεμία. Ε, η άλλη παρατήρηση για τον κατακαιρματισμό. Χρηματοπιστωτικό κατακαιρματισμό, ο οποίος επίσης η διασπορά έχει εξαφανιστεί σε μεγάλο βαθμό. Όταν ξεκινήσαμε είχαμε το υψηλότερο επίπεδο της διασπορά, του κατακαιρματισμού το 2012, Από το 2012 μέχρι τώρα είναι μειωτικέ οι τάσεις και παρατηρείται μια διαρκής βελτίωση σε χρηματοδοτήσεις, σε μείωσης του spread μεταξύ κρατών, διαφοράς επιτοκίων ε, μεταξύ κρατών και διατραπεζικών ε, δανεισμών και μεταξύ τομέων, δηλαδή είτε μεγαλύτερες είτε μικρότερες επιχειρήσεις. Οι δε τελευταίες μελέτες, μια πρόσφατη για διατραπεζικό διαλυσμό, δείχνει εξέλιξη αυτής της θετικής ε, τάσης και μάλιστα μια μελέτη που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η ίδια για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, η οποία μάλιστα μελέτη πριν απο δυο δύο-τρία χρόνια, όταν ρωτούσαν τις μικρομεσαίες ε, να εντοπίσουν το σοβαρότερο πρόβλημα που αντιμετώπιζαν πολύ συχνά, απαντούσαν τη δυσκολία προσέγγισης, ε, εξασφάλισης ε, πιστώσεως, ε, και αυτό πάλι με διαφορές ανάλογα με το είναι επαγγελματική δραστηριότητα ή την περιοχή. Τώρα η απάντηση είναι δεν μπορούμε να βρούμε πελάτες και η διαθεσιμότητα των κεφαλαίων των πιστώσεων ε, έρχονται τελευταία ως, ως πρόβλημα. Αντίστοιχα, και στη δική μας μελέτη όταν είχαμε ερώτημα για πρωταρχικό για πρωταρχική επιλογή και λόγους χορήγησης δανείου για τις τράπεζες, κριτήριο καλύτερα, η απάντηση ήταν ο κίνδυνος και βέβαια στην περιφέρεια ήταν πολύ ψηλότερος αυτός ο κίνδυνος από ό,τι στον πυρήνα και βέβαια όσο ήταν χαμηλότερες και οι ροές δανείων ε, στην περιφέρεια από ό,τι σε σχέση με, τον, ε, με το επίκεντρο. Ε, τώρα αυτό δεν εμφανίζεται καν ως κριτήριο ή μέλημα. Πρώτα εμφανίζεται η ζήτηση και μετά ο ανταγωνισμός για τις τράπεζες. Άρα και ασφαλώς είναι ικανοποιημένο το Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά νομίζω υπάρχουν ε, βάσιμοι λόγοι να είναι κανείς αισιόδοξο και ικανοποιημένο γιατί έχει οδηγήσει στον περιορισμό αυτή του κατακαιρματισμού η πολιτική μας. Ευχαριστώ κύριο Στάν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που ήρθατε. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι σίγουρα η νομισματική πολιτική ευθύνεται για την μακροχρηματοοικονομική σταθερότητα. Και θα, δεν θα πρέπει οι δημοσιονομικέ πολιτικέ να αντιβαίνουν στη νομισματική πολιτική. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε μια πρόσφατη πρόταση πρότεινε τον προσανατολισμό ε, στο δημοσιονομικό και πρότεινε χώρες όπως οι κατοχώρες ή η Γερμανία θα πρέπει να επενδύσουν περισσότερο, μέχρι 50 δισεκατομμύρια. Ε, και αυτό θα ήταν αντισυγκυριακή δημοσιονομική πολιτική. Τελικά, αυτό που έκανε η Υπουργό μα, ε, σήκωσε του ώμου τη και είπε δεν θα πρέπει καν να επεμβαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα, δεν θα έπρεπε καν να κάνει τέτοια σχόλια. Αυτό είναι όμω μια ευκαιρία που χάσαμε και που θα μπορούσε να συμβάλλει στη σταθεροποίηση στην Ευρωζώνη. Συμφωνείτε μαζί μου. Αυτή ήταν η πρώτη ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση, σχετικά να αφήσουμε την πρώτη. Φαίνεται ότι είστε από διαπομπέως ε, τράγος του Σόιμπλε. Σας ε, κατηγόρησε για την έξαρση του λαϊκισμού. Τώρα λέει το ευρώ είναι πολύ χαμηλά, σε χαμηλά επίπεδα για την Γερμανία. Μετά θα σας κατηγορήσει για υψηλό πληθωρισμό στη Γερμανία. Ξέρετε πόσο ευαίσθητη είναι η Γερμανία για τον πληθωρισμό. Για όλα εσείς Κάπω λοιπόν θα πρέπει να διαχειριστείτε τις διάφορες προσδοκίε, γιατί στόχο είναι να πλησιάσουμε το 2% πληθωρισμό, αλλά σε χώρες όπως η Γερμανία και η Ολλανδία ο πληθωρισμός θα είναι πολύ πάνω από το 2%. Τώρα για πόσο καιρό και τι θα συμβεί ε, και τι διαφορές ε, ε, πληθωρισμού θα προτιμούσατε. 1% μεταξύ Γερμανίας, Ολλανδίας και υπολείπων. Πάνω από 1% διαφορά στο επίπεδο πληθωρισμού. Τι θα προτιμούσατε. Ευχαριστώ. Δράγκη. Ω προ τη δεύτερη ερώτηση. Ας απαντήσω πρώτα στη δεύτερη σα ερώτηση. Καταρχήν οι διαφορές ε, στα ποσοστά πληθωρισμού δεν είναι κάτι καινούριο. Είχαμε ανέκαθεν τέτοιε διαφορές. Ακόμη και πριν από την κρίση και πολύ περισσότερο πριν από την κρίση είχαμε ε, αισθητέ διαφορές στα επίπεδα πληθωρισμού και διαφορέ υπάρχουν και σήμερα στα ποσοστά πληθωρισμού δικός μας στόχος ε, καθορίζεται ε, ως προς το ποσοστό πληθωρισμού για το σύνολο της Ευρωζώνης, όχι για τις μεμονωμένες χώρες. Τώρα, σε ό,τι αφορά διάφορες δηλώσεις, δεν θα σχολιάσω δηλώσεις ε, εθνικών πολιτικών, γιατί έγιναν πολλές δηλώσεις και δεν θα μπορούσα να τις σχολιάσω όλες. Πάντως, θυμάμαι τι είχε πει ο προκάτοχός μου, ο Βιμ Ντέιζενμπέρκ, ένας πολύ καλός Ολλανδός, όταν τον επέκριναν, για να μην πω όταν του επιτέθηκαν, για την νομισματική πολιτική που ακολουθούσε τότε η τράπεζα. Είχε πει πάνω κάτω ότι είναι κατανοητό για τους πολιτικούς, ιδιαίτερα σε προεκλογική περίοδο, να εκφέρουν τις απόψεις τους για την νομισματική πολιτική. Παρόλο που καλύτερα θα ήταν να έχουν μια ευγενική ανταλλαγή απόψεων από ότι να δακτυλοδεικνύουν κάποιου. Πάντως, είναι κατανοητό να εκφέρουν τι απόψει του οι πολιτικοί για την ε, νομισματική πολιτική, αλλά είναι επίση κατανοητό ανεξάρτητοι κεντρικοί τραπεζίτε να, να μην ακούν τέτοια σχόλια. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ε, τον δημοσιονομικό προσανατολισμό. Ε, δεν είναι σωστό αυτό που είπα ότι η νομισματική πολιτική είναι η μοναδική πολιτική. Είχαμε και εξαιρέσει. Μία εξαίρεση ήταν η Ολλανδία. Στην Ολλανδία εφαρμόστηκε και αποτελεσματική δημοσιονομική πολιτική από αυτήν την άποψη. Ε, και φορολογική πολιτική με ουσιώδεις τροποποίησης στην φορολογική νομοθεσία. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον δημοσιονομικό προσανατολισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο... Θεωρούμε σε γενικές γραμμές ότι ο σημερινός δημοσιονομικός προσανατολισμός είναι σωστός. Και μέχρι το τέλος του έτους ίσως τον κρίνουμε και ελαφρώς επεκτατικό αυτό τον προσανατολισμό, αυτή τη δημοσιονομική κατάσταση. Μερικέ χώρες μάλιστα αναβάθμισαν ε, τις δαπάνες του τα σχέδια δαπανών δεδομένη της μεταναστευτική κρίση ε, της ασφάλειας και των ε, πολυαριθμών αναγκών τους. Πάντως κατά κανόνα ο δημοσιονομικός προσανατολισμό ή η δημοσιονομική κατάσταση κάποιας χώρα θα πρέπει να αντανακλά φυσικά και την ανάγκη στήριξη τη ανάκαμψη, αλλά και την βιωσιμότητα της ανάκαμψη. Μίλησα προηγουμένω για χώρε που δεν έχουν δημοσιονομικό περιθώριο. Θα ήθελα τώρα να πω δύο λόγια για τι χώρε που έχουν τέτοιο δημοσιονομικό περιθώριο. Εδώ στην Ευρωζώνη έχουμε χώρε που έχουν δημοσιονομικό περιθώριο. Έχουν πλήρη απασχόληση. Και άλλε χώρε που δεν έχουν δημοσιονομικό περιθώριο και δεν έχουν πλήρη απασχόληση. Για τι δεύτερε είπα, σχολιάσα προηγουμένω, για, για την πρώτη κατηγορία χωρών, το να λέμε μια διάκριτη, ευρεία, δημοσιονομική επέκταση σε χώρες με πλήρη απασχόληση δεν έχει νόημα. Ίσως θα θέλαμε να χρησιμοποιηθεί αυτή η δυνατότητα, αυτός ο χώρος για την υπόλοιπη Ευρωζώνη. Αλλά δεν έχουμε σήμερα έναν άμεσο θεσμικό μηχανισμό ώστε έναν εθνικό δημοσιονομικό χώρο να το μετατρέπει η περιθώριο, να το μετατρέπει σε ευρωπαϊκό περιθώριο δημοσιονομικό της Ευρωζώνης. Οπότε, μέτρες δημοσιονομικές επεκτάσεις ίσως είναι θεμητές ε, οι εύλογες, αλλά θα πρέπει να ε, στοχεύουν στην αύξηση της ζήτησης και της παραγωγικότητας στις χώρες αυτές που τους ή άλλους έχουν πλήρη απασχόληση. Οπότε επενδύσεις στην παιδεία, στην ψηφιοποίηση, σε ειδικέ υποδομές θα ήταν σκόπιμες. Αλλά εγώ δεν θα ήμουν υπέρ ε, ευρείας δημοσιονομικής επέκτασης σε γενικές γραμμές. Ευχαριστώ. Ελπίζω να απάντησες σε ερωτήσεις. Γι' αυτό ε, μερικοί θεωρούμε ότι η δημοσιονομική ικανότητα της Ευρωζώνης ήταν ο μόνος τρόπος για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Περνάμε στο Κάτσι Διάη γρήγορα. Ζαριανόπουλος ε, πρώτα και μετά Κύρτσος. Ε, κύριε Τράκη, φαίνεται ότι οι διαπραγματεύσει για την αξιολόγηση του ελληνικού μνημονίου θα καταλήξουν. Φαίνεται ότι συμφωνείτε με την ελληνική κυβέρνηση για νέα μέτρα στους μισθούς, στι συντάξει στη μείωση του φορολόγιο του. Οπότε δεν θα σας ρωτήσω γι' αυτό. Θα σας ρωτήσω όμως για μια έκθεση της Ευρωπαϊκή Κεντρικής Τράπεζα που δημοσιεύθηκε τελευταία και που προωθεί, παύλα απαιτεί, αντικατάσταση των εργασιακών συμβάσεων σε επίπεδο κλάδου με εργασιακές συμβάσεις σε επίπεδο επιχείρησης για πιο ευέλικτους, άρα και πιο μικρούς μισθούς ακόμα. Ερώτηση, ερωτήσεις μάλλον. Σε τι τελικά αυτή η πολιτική ωφέλησε τους εργαζόμενους και τους εργοδότες είναι δεδομένο ότι ωφελήθηκαν, αφού και οι μισθοί μειώθηκαν και η ανεργία στην Ελλάδα παραμένει υψηλότατη και η ευέλικτη εργασία γενικεύεται όλο και περισσότερο με μισθούς τη τάξη των 200-250 ευρώ. Επειδή η ελληνική κυβέρνηση λέει ότι είναι καλή η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά κακό το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όσον αφορά το μισθολογικό και αυτό το ζήτημα, σε τι διαφέρει η άποψη Δούνου και Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η μείωση μισθών είναι εναλλακτική όσον αφορά τις ομαδικές απολύσεις που προωθούνται. Αυτή είναι η βέλτιστη πρακτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί πρόκειται περί εκβιασμού. Τέλος, πλεονάσματα υπάρχουν και μπορεί να βγουν και άλλα και να υπάρξει ανάκαμψη. Αλλά εδώ ακούμε ότι το πρώτο επιχείρημα ακόμα και σε ανάκαμψη είναι ότι δεν θα αυξηθούν οι μισθοί διότι θα ξαναγυρίσουμε πίσω στην κρίση. Τελικά, τελικό ερώτημα. Για ανάκαμψη όπως μιλάτε εσείς και η κυβέρνηση με σταθερότητα σημαίνει σαν προϋπόθεση απαραίτητη η μείωση των μισθών ώστε να προσελκυστούν ε, νέες επενδύσεις. Thank you, Ευχαριστώ κύριο Κίρτσος. Και άλλη ελληνική ερώτηση προς τον πρόεδρο Ντράγκη. Ε, γίνονται διαφορετικές εκτιμήσεις ως προς τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει καταλήξει πολύ αρνητικά συμπεράσματα ως προς τη βιωσιμότητα, ενώ ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας δείχνει μια συγκρατημένη ισοδοξία γι' αυτό. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Τι γνώμη έχει για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Καταλήξετε στο συμπέρασμα γι' αυτό. Πρόκειται να καταλήξετε σε σχετικό συμπέρασμα. Θα ακολουθήσετε τα ίδια κριτήρια, η διαφορετική προσέγγιση. Μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια. Thank you. I, unfortunately, Ευχαριστώ. Δυστυχώς. Έρχομαι στο πρώτο ερώτημα. Δεν γνωρίζω τι λέει η έκθεση του ΩΣΑ. Άρα μπορώ να σας απαντήσω, αλλά γραπτός αν το δέχεστε. I'm sorry? Yeah. Yeah. A written as European Central Bank. Θα σας δώσω γραπτή απάντηση ως Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για την έκθεση του ΩΣΑ, λέει ο κύριος Στράγκη. Το θέμα βέβαια είναι πως θα πρέπει να υπάρξουν μέτρα για την επιτάχυνση της απορρόφησης των ανέργων. Αυτό είναι σημαντικό. Τώρα, το είδος των μέτρων είναι κάτι το οποίο συζητείται στις διαπραγματεύσεις για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Κατά την άποψή μας, ε, και εδώ σχετίζεται και το άλλο σας ερώτημα ε, με αυτό, νομίζουμε ότι υπάρχει σημαντική πρόοδος που συντελείται στην Ελλάδα. Σημαντικές αλλαγές έχουν ήδη γίνει Τώρα, η ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης ε, κολλάει, αν θέλετε, λίγο πολύ στα εξής. Εκτιμάτε, πιστεύετε, καταρχάς, πως για να υπάρξει θετική αξιολόγηση της βιωσιμότητας του χρέους θα πρέπει να υπάρχει 3,5% πρωτογενές πλεόνασμα. Για αρκετά μακρά, δηλαδή χρονική περίοδο. Και αυτό είναι το ένα από τα σημεία στα οποία κολλάει διαπραγμάτευση. Το δεύτερο έχει να κάνει με, την, με το κλείσιμο του δημοσιονομικού χάσματος. Και το άλλο, κάποιες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, μεταξύ των οποίων μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, δικαστικό, ενέργεια, και θα πρόσθετα κι άλλη μία, άλλο ένα τομέα. Και εδώ μπορώ να μιλήσω για το ρόλο της ΕΚΤ. Είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό και αφορά την διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και πώς θα δοθεί νέα ε, δύναμη στο τραπεζικό σύστημα. Ο δικός μας ρόλος ε, της Τρόικας, θα τα τελευταία δύο-τρία χρόνια είναι ξεκάθαρη ότι αφορά το πιστοτικό τομέα που είναι και πιο κοντά αν θέλετε στις θεσμικές ε, εξουσίες και ικανότητες της ΕΚΤ και δυνατότητες. Σας ευχαριστώ πολύ. Για... Σας ευχαριστώ πολύ για τις πολύ ενδιαφέρουσες αυτές παρατηρήσεις. Είναι σημαντικός ο οικονομικός και νομισματικός διάλογος. Σημειώνω ιδιαίτερος τα όσα είπατε για τη σημασία του ρυθμιστικού πλαισίου που ορίζεται σε εθνικό επίπεδο. τα όσα ψηφίσαμε ως Επιτροπή για τη Βασιλεία διαφέρουν ιδιαίτερα από αυτά τα οποία μας είπε το Κογκρέσο και υπογραμμίσαμε στην επιστολή μας ότι υποστηρίζουμε υγιή και σωστά και εύρωστα πρότυπα. 29 Μαΐου είναι η προσεχής συνεδρίαση του διαλόγου. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία εδώ. Για colleagues. Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ. Έχω ανακοινώσει πριν περάσουμε στο επόμενο σημείο. Καταρχήν να σας υπενθυμίσω ότι ένα σεμινάριο μαζί με την budget για την χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων και τη σύνδεσή του με άλλα επενδυτικά ταμεία θα γίνει στις 8 Φεβρουαρίου, ημέρα Τετάρτη. Επίσης, η κοινή συνεδρίαση Econ Budget και ε, η κοινή συνεδρίαση και με την ε, Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού θα γίνει τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου στο Στρασβούργο των τριών επιτροπών κοινή συνεδρίαση. Κατά πάση πιθανότητα θα, θα ψηφίσουμε και όλα και τις εκθέσεις που αναβάλουμε αν δεν προλάβουμε σήμερα και θα έχουμε και την κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Προϋπολογισμών. Σημειώστε λοιπόν 13 Φεβρουαρίου σημαντική κοινή συνεδρίαση ε, στο Στρασβούργο. Διορθωτικό ΜΥΦΙΤ 2. Έχουν κυκλοφορήσει μεταφράσεις του διορθωτικού ε, στις 31 Ιανουαρίου για το ΜΥΦΙΤ 2. Το διορθωτικό το ετοίμασαν οι γλωσσομαθείς νομικοί και παραπέμφθηκε στην ΕΚΟΝ που είναι αρμόδια κατορουσία επιτροπή με βάση το άρθρο 231 και σε περίπτωση που δεν υποβληθούν ενστάσει από την Επιτροπή, το διορθωτικό για το MIFID 2 θα υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ανακοινωθεί στην Ολομέλεια κατά πάσα πιθανότητα στη δεύτερη Ολομέλεια του Φεβρουαρίου και θα θεωρηθεί ότι εγκρίνεται εκτός και αν, αντι... αν ισχύσει το 176 και κάποιες ομάδες αντιταχθούν στο διορθωτικό αυτό με βάση το απαραίτητο αριθμό ψήφων και ευρωβουλευτών που χρειάζονται. Έχουμε γνωμοδότηση τώρα για το 290-291 αυτό αφορά το Προεδρείο, Οικονομική Διακυβέρνηση, Συντονιστές της Επιτροπής Εκο... Αυτό το συμφώνησαν ούτως ή άλλως έκτακτη κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή ε, Προπολογισμών. Θα λάβει χώρα στο Στρασβούργο παρουσία του Αντιπρόεδρου Κατάινεν. Η μελλοντική διαρθρωτική διάλογη. Ευρωπαϊκό εξάμεινο Ντομπρόφσκι και Μοσκοβισή. Χρηματοοικονομικές υπηρεσίε Ντομπρόφσκι ε, Φορολογία Μοσκοβισή. Ανταλλαγή απόψε με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου και με μέλη άλλων ε, συμβουλίων θα γίνει στην ΕΚΟΝ αλλά δεν ξέρουμε ακόμα πότε, θα σας το ανακοινώσουμε όταν καταλήξουμε. Επίσης ε, θα στείλουμε επιστολή στον πρόεδρο του, ΕΛΚ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζητώντας επιστολή προς την Εστονική Προεδρία για να αλλάξει ε, το άρθρο 13 για την οικονομική διακυβέρνηση που θα γίνει στο Τάλιν ε, στην Πράσινη Εβδομάδα, να αλλάξει ημερομηνία. Επίσης θα έχουμε μια συνεδρίαση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Συνεργασίας κατά πάσα πιθανότητα 15 Φεβρουαρίου θα συζητηθούν θέματα και αγοράς εργασίας. Επίσης, νέα διερευνητική αποστολή θα γίνει στην Ελλάδα. Η ομάδα εργασίας θα ασχοληθεί με τις χώρες που έχουν εξέλθει από προγράμματα διάσωσης, παρουσία πυρογνωμόνων και ε, μη κυβερνητικών οργανώσεων. Επίσης, ότι το τον πρώην πρόεδρο της ε, Ελστάτ, ε, θα γίνει ε, θα γίνουν τέσσερι συνεδριάσει και μία παρουσία του Επιτρόπου Μεσκοβίση το Μάρτιο. Επίση, οι Υπουργοί Οικονομικών των, μεγαλύτερων, τεσσάρων μεγαλύτερων χωρών θα συζητήσουν το θέμα τη Ελλάδα. μεταρρυθμίσεις αγορά εργασία, παρουσία και Ελλήνων Υπουργών, κατάσταση του Εθνικού Ταμείου Αποκρατικοποιήσεων και τέλος έλεγχος για, τον, για τις πράξεις για 21 για, την, για τα κανονιστικά στάνταρ του MIFID. Ξεκίνησε η διαδικασία αντιρρήσεως στην ΕΚΟΝ και οι πολιτικές ομάδες που θέλουν να το επισημάνουν μπορούν να το κάνουν και στην Ολομέλεια. Ε, ο πρόεδρος ε, επιβεβαίωσε την ε, ανακοίνωση που έγινε από τον πρόεδρο Ταγιάννη και θα ήθελα να ζητήσω από τις ομάδες να βρούμε κάποια λύση για να ολοκληρωθεί η εκλογή των μελών του Προεδρείου μας. Γιατί με τον ε, Μάρκος νιώθουμε μοναξιά. Έχουμε θέσεις αντιπροέδρων ελεύθερες που πρέπει να πληρωθούν. Και περνάμε στο σημείο, στα σημεία 6, 7 και 8 της ημερήσιας διάταξης, στην απαλλαγή των τριών αρχών. Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων και Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών. Ο εισηγητής μας είναι ο κύριος Άντερ Λούνς. Θα εξετάσουμε τις τροπολογίες. Παρακαλώ, εισηγητής. Ευχαριστώ και συντομία θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους συναδέλφους που, βρήκαν το χρόνο και συνέταξαν πολύ αξιόλογες τροπολογίες. Θα τις εξετάσουμε τώρα κατά την εξέταση των συμβαστικών προτάσεων και ευελπιστώ ότι θα συντάξω και θα μοιράσω μέχρι την Τετάρτη τις συμβαστικές αυτές τροπολογίες, το αργότερο Τετάρτη το απόγευμα και όπως συνέβη και την τελευταία διετία, πρόταση είναι να μην συνεδριάσουν οι σκιώδει ηγητέ, αλλά να ακολουθήσουμε τη γραπτή διαδικασία για την εξέταση των συμβαστικών τροπολογιών. Σήμερα να σταθώ σε δύο μόνο σημεία. Κάποιες ομάδες στην Επιτροπή υπέβαλαν μια πλειάδα θεμάτων ε, και στις τροπολογίες τους αναφέρθηκαν μερικές ομάδες στην αλλογικότητα, άλλες στην προστασία καταναλωτή, σε διαφάνεια και ούτω καθεξής. Πάντως είμαι πεπισμένος ότι θα καταφέρουμε να συνδυάσουμε αυτές τις τροπολογίες και θα τις καλύψουμε στις συμβαστικές τροπολογίες. Δεύτερον, να πω δύο λόγια για δύο τροπολογίες, τις 26 ε, και 33 της Επιτροπής για την ε, Αρχή για τις Τράπεζες, τροπολογίες Λάγκεν και Κάρας και οι δύο αφορούν τη δυνατότητα συμπερίληψης της ΕΑΤ στο σύστημα εποπτείας ε, των τραπεζών της ΕΚΤ. Και μάλιστα ο κύριος Κάρας αναφέρει τη δυνατότητα να συμπεριληφθεί η ΕΑΤ στον ε, ενιαίο εποπτικό μηχανισμό στη Φραγκφούρτη. Και μια και θα, θεωρθεί, εξεταστεί το θέμα της ΕΑΤ, ούτως ή άλλως δεν νομίζω ότι η γνωμοδότηση μόνο η κατάλληλη ευκαιρία γι' αυτό. Μερικοί θέλουν η Άτη να μεταφερθεί στη Φραγκφούρτη. Και, φαντα... και... Α, ο κύριο Χέι και άλλοι θα προτιμούσαν να, να μετακομίσει στη... στο Δουβλίνο. Φαντάζομαι άλλοι θα ήθελαν την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών στο Μιλάνο. Δεν νομίζω να, φροντίσει, να ζητήσει κάποιο να έρθει στι Βρυξέλλε. Βέβαια, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Πάντω, στην συμβαστική τροπολογία θα πούμε κάτι γενικό να εξασφαλίσει τη διαφάνεια, τη μέγιστη διαφάνεια στη διαδικασία λήψη αποφάσεων σε σχέση με τη μελλοντική έδρα της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών. Αυτά και περιμένω τις απόψεις των σχεδόν εισηγητών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Πολύ σωστό αυτό που είπατε βεβαίω. Δεν είναι η ώρα, η θέση για τέτοια συζήτηση στην έκθεση περί απαλλαγής. Ούτε για τις συνέπειες ε, της, εκ, της αποφάσης για το Brexit, ούτε η κατανομή των ε, εδρών όπως τη ΣΕΑΤ. Κύριε Λάγκα, εκ του ΕΛΚΑ. Κοιτάξτε, εν όλο έχουμε περί 100 τροπολογίες για τις τρεις εκθέσεις απαλλαγής, αν το μετράω σωστά. οι οποίες ε, μάλιστα τροπολογίες είναι λίγο πολύ ε, οπότε δεν νομίζω θα έχει πρόβλημα στην υποστήριξη που θα δοθεί στον εισηγητή. Ένα-δύο μόνο ζητήματα θέλω να επισημάνω. Πρώτον, ε, οι πόροι, με τις ε, επιφυλάξεις που εκφράζονται προς τις περικοπές των πόρων μετακύληση πόρων είναι το ελάχιστο ή μη τι άλλο για την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής ε, ε, υποστήριξης δεδομένων και των νέων νομοθετικών αρμοδιοτήτων. Επίσης, έχει ζητήσει η έκθεση Φέρμπερ να τηρηθούν αυστηρά οι όροι των εντολών αυτών των υπηρεσιών. Το υποστηρίζει βέβαια απερίφραστα το ολόκληρο το έλκος ομάδα, η εντολή για την, αρχή, για την ασφαλιστική αρχή βλέπουμε ότι έχει μάλλον υπερβληθεί. Ιδιαίτερα για την ασφαλιστική αρχή για την ε, αρχή εποπτείας χρηματοπιστωτικών αγορών ο συνάδελφος Κουντουλίτσια έχει, έχει επικρίνει τις αντίστοιχες ε, δραστηριότητες της Ρουμανικής Αρχής. Και νομίζω ότι όχι μόνο αυτός αλλά και άλλοι επισημαίνουν ότι δεν λειτουργεί σωστά η ασφαλιστική αρχή. Άρα μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να γίνει συζήτηση επί της ε, ουσίας των, ε, της διατύπωσης για την ε, μετάβαση στη Φραγκφούρτη. που θα μπορούσε να προχωρήσει όταν ολοκληρωθεί το Brexit. Ναι, δεν πρέπει να μας απασχολήσει τώρα, αλλά πάντως πρέπει να μας, να μας απασχολήσει η συνάφεια με τον SSM. Και η ΕΑΤ, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, έχει έως το 2026 επιφορτιστεί με ένα, με ένα μισθωτήριο συμβόλαιο που ως εκ τούτου σημαίνει σημαντική επιβάρυνση και των οικονομικών της. Το που θα εγκατασταθεί στη συνέχεια δεν έχει μεγάλη σημασία. Πολλοί είναι αυτοί που ε, ενδιαφέρονται, το ξέρουμε. Θα, έχει, θα ληφθεί η απόφαση με όρους πολιτικούς ασφαλώς. Ε, αλλά ιδιαίτερη σημασία έχουν ε, αυτές οι επιφυλάξεις. Επίσης, Γκίγκολ, Τσάνι, Μαριάς και άλλοι έχουν ε, κάνει τις επισημάνσεις τους. Ο κύριος Γκίγκολτ ζητά, ζητεί να υπάρξει μια διευκόλυνση για τους καταγγέλλοντες υπαλλήλου και για την ΕΑΤ. Και γενικά νομίζω ότι αυτό είναι μια πρόταση που θα πρέπει να μπει σε, μια πρώτη, ε, σε έναν πρώτο απολογισμό δραστηριοτήτων και για τις τρεις αρχές. Να τα προβλήματα επιτοπλίστων έχουν επιληθεί. Καλώς ευχαριστώ, σοσιαλιστές δημοκράτες εκ μέρους του κύριου Φουντσουλικά. Ο κύριος Περί... Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα λυπούμε που δεν μπορεί να είναι εδώ και ο εισηγητής. Ο κύριος Φουντσουλικά ζητά και αυτό συγγνώμη. Όμως τον αντικαθιστώ εγώ και θα ήθελα να σας πω ότι οι τρεις αυτές αρχές σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικές και σε ό,τι αφορά την αιτήσια απαλλαγή θεωρούμε ότι αυτή είναι μια ευκαιρία για να εντοπίσουμε κάποια προβλήματα. Η βασική μας ανησυχία είναι να εξασφαλιστεί ότι εν λόγω αρχές θα έχουν επαρκείς πόρους ώστε να μπορούν να, να φέρουν σε πέρα στα καθήκοντά τους ανεξάρτητα και αποτελεσματικά. Και από τη δική μας οπτική γωνία, επέκταση των καθηκόντων των αρχών αυτών θα πρέπει να ε, συνοδεύεται και από αύξηση των πόρων και εξορθολογισμό των ήδη υφιστάμενων. Θα ήθελα επίση να υπογραμμίσω ότι οι τροπολογίε που έχουμε καταθέσει ω ομάδα, ιδίω για τι παραγράφου 2 και 4, θα ληφθούν, ελπίζω, από τον εισηγητή. Έτσι πιστεύω. Και ό,τι αφορά τη γραπτή διαδικασία που πρότεινε ο εισηγητή, νομίζω ότι είναι ένα λόγο για να έχουμε ακόμη μεγαλύτερη ισοδοξία για το ενδεχόμενο καλών συμβιβαστικών προτάσεων που θα δισκεδάσουν τις ανησυχίες που εκφράζει η ομάδα μας, που έχει εκφράσει η ομάδα μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η ECR έχει κάποιο πρόσωπο εδώ. Α, τι λέω, είστε εσείς ε, ο εισηγητής από το ECR, ναι, με συγχωρείτε. Άλντε, ο κύριος Τόρβαλτς. Ε, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. στα γραπτά μου σχόλια ε, είχα περιλάβει και κάποια κάπως πιο, πώς να διπλωματικά σχόλια για ορισμένες από τις τροπολογίες. Αλλά ο ε, πολύ ξεκάθαρα παρουσίασε την απόψη του για σαν λόγο τροπολογίας οπότε εγώ νομίζω ότι δεν χρειάζεται να σχολιάσω καν. Συμφωνώ και θα προσπαθήσω με τεκμηριωμένο τρόπο να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με ομαλό τρόπο. Σε ό,τι αφορά τώρα την έκθεση, είναι καλή, ισορροπημένη, σε καλό ύφος είναι γραμμένη και ελπίζω ότι παρά ορισμένες τροπολογίες θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε και να προχωρήσουμε. Επίκειται άλλωστε η ε, πανεξέταση και αναθεώρηση αυτών των αρχών. Οπότε φαντάζομαι ότι θα τα δούμε πιο λεπτομεριακά τότε. Προσβλέπω λοιπόν στην καλή συνεργασία με τον εισηγητή, τους λοιπούς σκιώδεις και δεν βλέπω να υπάρχει κάποιο πραγματικό πρόβλημα στον ορίζοντα. Thank you. Ευχαριστώ. Κανείς από την ΚΟΕ ο Σβέν από τους Πράσινους. Αγαπητοί συνάδελφοι, να ευχαριστήσω καταρχάς τον εισηγητή μας για την ε, σαφή και εξόλογη γνωμοδότησή του, με την οποία συμφωνούμε σε πολλά σημεία. Κυρίως με την πρόταση να αλλάξει το χρηματοδοτικό καθεστώς και να συμπεριληφθεί και η αναλογικότητα. Επίσης, να βελτιωθεί η ποιότητα και η διαφάνεια σε ό,τι αφορά τα πρακτικά των συναντήσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Όλα αυτά μας βρίσκουν απόλυτα σύμφωνος και είναι πολύ σημαντικά θέματα. Επίσης, ευχαριστώ και τον κύριο Βέρνερ Λάγκεν που συμφώνησε με την πρωτοβουλία μας να συμπεριληφθεί και η προστασία των καταγγελόντων, των whistleblowers θα πρέπει να ε, προβληθεί καλύτερα αυτό το θέμα. Ε, και καλό θα ήταν να το συμπεριλάβουμε εδώ. Άλλωστε και στο παρελθόν ε, είχαμε κάποια κοινή προσπάθεια για το σημείο αυτό. Τώρα, πού διαφωνούμε. Υπάρχει εδώ κέριο θέμα κατά τη γνώμη μου και μερικές τροπολογίες, όπως είπε Βένερ Λάγκεν, αμφισβητούν το, αμφισβητούν το κατά πόσο οι αρχές αυτές και κυρίως η ασφαλιστική αρχή και η αρχή επαγγελματικών συντάξεων πληρώνουν την εντολή τους. Έχω την αίσθηση, όπως και άλλοι συνάδελφοι, ότι έχουν υπερβεί την εντολή τους. Και προσοχή λοιπόν όμως σε μια απαλλαγή, σε μια έκθεση απαλλαγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να περιλαμβάνουμε τέτοιες δηλώσει περί καταστρατήγηση ή υπέρβασης της εντολή. Για να κάνουμε τέτοιου τέτοιους και να απευθύνουμε τέτοιε κατηγορίες θα πρέπει να έχουμε πρώτα ε, συγκεντρώσει τεκμήρια που να συνηγορούν υπέρ αυτής της άποψη. Επίσης αυτές οι αρχές, όπω είπε και ο εισηγητή, έχουν κάποιες ε, μη βασικέ δραστηριότητε. Ε, στην παράγραφο 3 ε, θα πρέπει καταρχήν να λάβουμε υπόψη ότι η εντολή περιλαμβάνει την προστασία του καταναλωτή, την προστασία του επενδυτή και κάποια θέματα ε, χρηματοοικονομικής σταθερότητας. Οπότε είναι σημαντικές αυτές οι εντολές τους και Μάλιστα σε μερικές περιπτώσεις αυτές οι αρχές δεν μπόρεσαν να ε, εκπληρώσουν την εντολή τους γιατί οι αρμόδιες αρχές των εθνικών μελών δεν έδιναν στην αρχή αυτή την πραγματική αρμοδιότητα για δράση, παρόλο που η εντολή το προέβλεπε. Αυτό επισημαίνουμε σε μερικές τροπολογίες. Ε, εγώ δεν συμφωνώ ότι υπερέβησαν τις εντολές τους οι αρχές αυτές. Εγώ θα έλεγα ότι υπήρχαν κάποια προβλήματα αναλογικότητα σε μερικές περιπτώσεις και σε αυτό συμφωνούμε ότι σε μερικές περιπτώσεις θεσπίστηκαν κανόνες που ήταν υπερβολικές ό,τι αφορά την επιβάρηση στους μικρούς τελεστές της αγοράς, αλλά δύσκολο είναι να βρούμε περιπτώσεις όπου μπόρεσαν οι αρχές να εκπληρώσουν πλήρως την εντολή τους. Και μάλιστα σε μία τροπολογία μας επισημαίνουμε μία σειρά θεμάτων στα οποία δεν κατάφεραν οι αρχές να υλοποιήσουν την εντολή τους. Και μάλιστα ε, εδώ υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ των πολιτικών ομάδων. Οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες υπενήχθηκαν την προστασία του καταναλωτή. Φαίνεται ότι συμφωνούμε μάλλον ως προς το θέμα αυτό. Πάντως ε, το ζήτημα αυτό είναι ευαίσθητο και θα φανεί και στις τροπολογίες. Το μόνο πρόβλημα που έχουμε θέμα ουσίας είναι αυτό. Το θέμα είναι το θέμα της έδρας. Εκεί πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε μια λογική συμβαστική τροπολογία. Αν και το Κοινοβούλιο ήταν υπέρ μια ενιαία έδρας, προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα αυτών των αρχών. Και κάτι τέτοιο θα είχε νόημα να το συνεχίσουμε. Αυτό που δεν καταλαβαίνω και θα ήθελα να ρωτήσω του Σλάγκερ και Κάρας για διευκρίνηση. Είπατε να μπει η ΕΑΤ στον νέο αποπτικό μηχανισμό. Θέλετε, δηλαδή στην ΕΚΤ ουσιαστικά, θέλετε να αυξηθούν ακόμη περισσότερο οι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή μήπως καλύτερα να ζητήσουμε έναν εξωτερικό επόπτη εκτός της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που θα περιλαμβάνει και τις λειτουργίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών στην εποπτεία του. Αλλά το να ζητήσουμε να περιληφθεί αυτή η λειτουργία στο πλαίσιο της ΕΚΤ, ουσιαστικά αποδυναμώνοντας τον δημοκρατικό έλεγχο, δεν είμαι σίγουρος ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συμφωνήσει με μια τέτοια προσέγγιση. Ευχαριστώ. Η ΕΝΕΦ. Όχι. Άλλες ομάδε δεν βλέπω. Κύριος Λάγκεν, πολύ στόμα. Άλλο υπέρβαση εντολή σε πρώτη γραμμή έχει να κάνει με την πρωτοβάθμια νομοθεσία και τα σχετικά νομοθετήματα. Πρέπει να παραμείνουν λοιπόν να περιοριστούν στο level 1, στο πρώτο επίπεδο, οι αρχές και να μην το υπερβούν. Μπορούμε να δούμε όλα αυτά βέβαια στην ε, έρευνα, στην αναθεώρηση. Δεύτερον, Κάνω την ε, τροπολογία για την ενοποίηση, για την ολοκλήρωση, όχι γιατί θεωρώ ότι είναι απαραίτητα, αλλά γιατί η τραπεζική εποπτεία και τα νομισματικά θα πρέπει κάποια στιγμή να φύγουν από τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και να διαχωριστούν. Και δεν θέλω να είναι δύο παράλληλοι οργανισμοί αρμόδιοι για τα θέματα αυτά. Ο εισηγητής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους τους εισηγητές για τις παρατηρήσεις τους. Όπως υπόθηκε, νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε στις τρεις αυτές νομοδοτήσεις, να τις ε, διευκρινίσουμε στο μέγιστο δυνατό, αλλά για να τις κάνουμε και πιο σύντομα. Σύντομες. Για τους πόρους, καταρχάς το σχόλιο του κυρίου Λάγκεν αλλά και των ε, Σοσιαλιστών Δημοκρατών και του Σβέν Γκίγκολτ. Πρέπει να μπορούν να εκτελούν το έργο τους, το εποπτικό. Η εντολή δεύτερον προβλέπεται στις συμβαστικές προτάσεις για Τετάρτη το αργότερο. Την ανάγκη της ε, νομιμότητας προσπαθούμε να καλύψουμε για την ΕΑΤ. κύριε Λάγκεν. Μερικές πληροφορίες φαίνεται ότι έχουν εισαγαγή ρήτρα ε, υπαναχώρησης που μπορεί να ενεργοποιηθεί το 2020. Η διάρρηξη της σύμβασης. Επομένως ε, δεν υπάρχει ζήτημα σε σχέση με το μισθωτήριο. Η ομάδα μας κάνει ένα σεμινάριο αργότερα το Φεβρουάριο. Σας το λέω να έρθετε. Σβέν, το τελευταίο. Για τη διαφάνεια. Θα προβλεφθεί στις ε, συμβαστικές τροπολογίες. και τα ζητήματα που θεωρούνται ε, όχι κεντρικά, ε, θα καλυφθούν τους άλλους μαζί με τις αρχές της αναλογικότητας κτλ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Η ψηφοφορία λαμβάνει χώρα στις 27 Φεβρουαρίου και 23 Μαρτίου για την Επιτροπή των του Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Υπογραμμίζω τα λόγια του κυρίου Λόγια. της υπέρβασης του πλαίσιου αρμοδιοτήτων. Έχουμε εμείς ένα ισχυρό εργαλείο στα χέρια μας. Και μπορούμε να εξετάσουμε όχι μόνο πώς εφαρμόζεται, πώς επιτελούν την εντολή τους, αλλά και αν τηρούν τα ωριά της με, με την υποπτία μας. Κύριος Λάγκεν εκτός μικροφώνου δεν ακούγεται. Μα είναι, είναι ισχυρό, ισχυρό εργαλείο και πάντα βεβαίως προτιμότερη η πρόληψη και ξέρουμε ότι μπορείς, μπορείτε εσείς προληπτικά να έχετε πολύ καλή δράση, αλλά υπάρχει και το άλλο, η άλλη δυνατότητα. Και μην ξεχνάμε τις διαφορές μεταξύ φορέων της ε, Ευρωζώνης και φορέων που εποπτεύουν τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά, αλλά όπως είπαμε θα γίνει και αναθεώρηση της δράσεως των υπηρεσιών όπου και θα συζητηθούν όλα αυτά τα ζητήματα. Σας ευχαριστώ θερμά. Πολύ ενδιαφέρουσα η συνεδρίαση. Ολοκληρώνουμε έτσι τη συνεδρίασή μας. Η προσεχής Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 7 το βράδυ.